Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, bonjour σε όλους. Good afternoon. Good afternoon. Καλώς ορίσατε σε αυτήν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας που όπως συνήθως έχει πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Πολλά σημεία, πάρα πολλά σημεία. Και ένα επιπλέον θέμα με την πολωνική αντιπροσωπή από το Κοινοβούλιο από τις 18.30 ε, ε, μέχρι τις 19.30. 6.30 Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Οπότε, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Τα σημεία 5 και 6 που έχουν να κάνουν με την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και Νορβηγίας για τη διαδικασία ε, την διαδικαστική συνδρομή και παράδοση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναβληθεί. Αν αυτόν όμω, έχουμε βάλει ένα σημείο. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρώμα. Η κυρία Λίδια Γερόκα είναι η συγκήτρια που σήμερα το απόγευμα θα μας παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων και το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά αυτήν την τόσο λεπτή και ευαίσθητη έκθεση. Εφόσον συμφωνείτε, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 2, που είναι οι ανακοινώσει του Πρόεδρου. In these announcements, I suggest we endorse εγκρίνουμε τις αποφάσεις του, των συντονιστών για, την, για τους εξής εισηγητές. Η κυρία Ντέβορα Σερακιάνη, πρόταση προκειμένου η Κροατία να συμμετέχει στο παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά. Δεύτερον, η κυρία Σόνια Αλφάνο, η συγκίτρια για έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, ο κύριος Ντένις Δε Γιόγκ, έκθεση πρωτοβουλίας για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ποινικό δίκαιο, εγκληματικό δίκαιο. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν έχει ακόμα δώσει την απόφασή της επ' αυτών. Είναι σε κρεμότητα δηλαδή αυτό το θέμα. Συμφωνείτε λοιπόν μετά την ε, συνάντηση των συντονιστών είχαμε αυτές τις συστάσεις. Εφόσον συμφωνείτε, εγκρίνονται από μας. Στα τέλη τώρα της ε, τακτικής αυτής της συνεδρίασης θα συναντηθούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Πολωνικού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσουμε για την Πολωνική Προεδρία Και θα ήθελα να θίξουμε και μερικά πράγματα, όπως είναι το TFTP, όπως επίσης και την Europol και την Eurojust και πώς λογοδοτούν τα σώματα αυτά σε μας. Ως πρόεδρος λοιπόν σας προσκαλώ όλους στην συνάντηση αυτή, η οποία θα λάβει η χώρα γύρω στις 6 και 30 σήμερα. Θα κρατήσει μία ώρα περίπου. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη τώρα, έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων που είχαμε. Συμφωνείτε? εγκρίνονται τα πρακτικά. Οπότε ξεκινάμε τώρα με την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, σας υπενθυμίζω. Φροντίστε να έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί για να μπορέσετε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τι, την ξεχάσατε? Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα κύριε Άλβαρο. Ε, τι να κάνω, πρέπει να σηκώσω το χέρι μου κάθε φορά. Τι να κάνω, Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εντάξει, θα υπολογίσουμε την ψήφο σου. Αλλά κρίμα. Για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα πρόκειται για τον Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Μεγάλων Πληροφοριακών Συστημάτων. Και ξεχνάτε την ηλεκτρική σας κάρτα. Εισηγητής ο κύριος Κάρλος Κόγιο. ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης, ενδεικτική ψηφοφορία, αλλά προηγουμένως ίσως ο κύριος Κοέγιο να θέλει να πάρει το λόγο για να μας εξηγήσει λίγο την έκθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδες εισηγητέ και όλους τους συναδέρφους που υπέβαλαν ε, τροπολογίες και συμφώνησαν με τις συμβιβαστικές που ετοιμάσαμε μαζί. Χωρί τη στήριξή τους και χωρί τη δικιά τους δουλειά δεν θα ήταν δυνατόν σήμερα να έχουμε σε αυτό το στάδιο το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Συνένεση δηλαδή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δεύτερον, θέλω να πω ότι θλίβομαι που δεν υπάρχει συμφωνία με την προφορική τροπολογία του Άλβαρο. Συνήθω συμφωνώ με τι τροπολογίε του. Είναι καλές, πολύ σωστές και πολύ καλά διατυπωμένες. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι από την αρχή δεν θα έπρεπε αυτό το θέμα να αποτελήσει μήλο της ε, έρηδος μεταξύ των χωρών μελών. Και γι' αυτό και πρότεινα να βάλουμε ένα άρθρο με τα κριτήριά μας. Και εφόσον το Συμβούλιο ακολουθήσει τα κριτήριά μας και καταλήξει σε συμπέρασμα, σε απόφαση, εμείς δεν θα έπρεπε να αντισταθούμε σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου. Τώρα η προφορική τροπολογία του Αλεξάνδρου Άλβαρο, ακόμα και αν είναι στα σκεπτικά, δίνει μια προτίμηση στην Εστονία σε σχέση με τη Γαλλία. Και κατά τη γνώμη μου εμείς θα έπρεπε να κρατήσουμε μια ουδέτερη θέση όσον αφορά την τοποθεσία που θα είναι δηλαδή ο οργανισμός. Λυπάμαι λοιπόν που διαφωνώ μαζί σου αυτή τη φορά Άλβαρο, αλλά είμαι υποχρεωμένο να ζητήσω από τους συναδέλφους να καταψυχηθήσουν την προφορική σου τροπολογία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε τον εισηγητή τον κύριο Κοέγιο. Η κυρία Σιλβίκη Γιόμ, και ο ε, εισηγήτρια Α, όχι, απλώς ευχαριστώ λέμε. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη δουλειά αυτή. Άλλος κανείς θέλει το λόγο εδώ κάτι να προσθέσει, η Επιτροπή μήπως. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Ξεκινάει η ψηφοφορία και ξεκινάμε με την τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά.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 53. Όχι. καλύτερα από την ανέα. Ωραία. 54 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία αριθμός 1, κοντ, υπέρ. Against. Αποχές, απορρίφθηκε. Συμβαστική αριθμός 3, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Κοντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 20 και 63 γιατί είναι ίδιες με προστίκη. 20-63, μαζί τις ψηφίζουμε. 20 και 63, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 και 64 τώρα. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρόεδρε, 28, 29 και 30 μπορούμε να τις ψηφίσουμε και τις τρεις μαζί. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Συμφωνείτε μαζί. Τις ψηφίζουμε και τι τρει υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνονται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε μαζί και τη 10, 11, 12, 5 και 13. λέει ο βουλευτής. Ε, συμφωνείτε, λέει ο πρόεδρος. Τι, διαδικαστικό, δεν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. μια, στιγμή, μια στιγμή να γυρίσω το κουμπί να βρω τη μετάφραση, λέει ο πρόεδρος. Τώρα μπορείτε να μιλήσετε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα τη 13 να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Τα υπόλοιπα εντάξει. απορρίπτεται για την 13. Οπότε ψηφίζουμε τις υπόλοιπες από τον μπλοκ μαζί, τις τροπολογίες, χωρίς τη 13 όμως. 10, 11, 12 και 5 μαζί. Έτσι, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τώρα τη 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε, τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 73. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, 35 και 36 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Πρόεδρο έχει κάνει αντίρρηση. Ωραία, ε, τι ψηφίζουμε μαζί λοιπόν. 34, 35 και 36. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 και 18 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 και 80 μαζί για την ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Πρόεδρε, συγγνώμη. Μπορείτε παρακαλώ να δείτε από την 19 μέχρι την 23. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε αν μπλοκ όλες μαζί. Και την 19, 20, 22, 23. 19, 20, 22, 23, 21, 22, 23. Όλες αυτές μαζί είπατε, έτσι. Υπάρχει καμιά αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 24 τώρα προπολογίζουν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 κοντ ελέγχου προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Extensions. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Ελέγχου προπολογισμού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα σκεπτικά. Τροπολογία αριθμός 1 προπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του κύριου Άλβαρο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 45. Ξεκινάει η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 16 υπέρ, 15 κατά. Δεν δούλεψε το μηχάνημά σας, ρωτάει ο πρόεδρος. Κάποιον παρεμβαίνει ή κάνατε λάθος. Α, πρέπει να μετρήσουμε τον κύριο Άλβαρο που ψηφίζει υπέρ, έτσι δεν είναι. Άρα είναι 16-16. Τότε τι κάνουμε, λέει ο πρόεδρος. Your vote is against. So yes, I say. But Mr. Alvaro, Mr. 17 to 16, eh? 16-16 είναι το αποτέλεσμα. Ε. Τι κάνουμε? Κοιτάξτε, προσθέτω μία ψήφο υπέρ που είναι του κύριου Άλβαρο και άλλη μία κατά για την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Οπότε είναι 16-15. Μα και 16-16 να είναι, λέει κάποιο από την αίθουσα, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε και πάλι. Καλά, θα ελέγξουμε και πάλι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 45. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Now the vote is, <laughs> Now the vote is closed. I'm so sorry, Sophie. <laughs> so, now it's Λοιπόν, το αποτέλεσμα τώρα είναι 16-16. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. Κύριε Άλβαρο, έτσι απορρίπτεται. Και πάμε στην τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 2 προϋπολογισμών τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 τώρα προπολογισμών υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 προπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και 41. Τελευταία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, έτσι. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας 29 υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Συνεπώς η έκθεση εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον κύριο Κάρλος Κοέγιο. Συγγνώμη, συγγνώμη εδώ, πρόεδρε. Κατά λάθο καταψήφισα, ενώ ήθελα να υπερψηφίσω. Το λέω για να διορθωθεί παρακαλώ στα πρακτικά και συγγνώμη για το λάθος που έκανα. Μπορούμε να το κάνουμε, άρα έχουμε άλλη μία ψήφο υπέρ και μία λιγότερη στα κατά. Καλώς, ωραία. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή και όλους σας. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μεσής διάταξης. Said, having postponed the agreement on Iceland and... Και όπως σας είπα, μια που αναβάλουμε τη συζήτηση των θεμάτων της και Νορβηγία, θα περάσουμε σε ένα καινούριο θέμα που είναι η της Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη των Ρώμα στις κοινωνίες. Υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο. Και θα ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Λίβια Γερόκα, που θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασία του θέματος. Περιμένουμε να γίνει μια βελέτη, που θα παρουσιαστεί προσεχώς. Και τα προσωρινά συμπεράσματα θα έχουμε στις 26 Οκτωβρίου, στην επόμενη μας συνεδρίαση της Λίμπη. Κύριε Λίβια Γιαρόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα έργο εργασία που, έχει, που δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στα γερμανικά και στα γαλλικά όπως περιμέναμε. Οι μεταφράσει αυτέ που δυστυχώ δεν είναι ακόμα έτοιμε, από όσοι μου λέμε, θα είναι έτοιμε στι 15 Οκτωβρίου. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, εάν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στις 26 Οκτωβρίου για μισή ώρα, όταν θα ακούσουμε την έκθεση των προσωρινών αποτελεσμάτων της μελέτης. Μόλις έχουμε λοιπόν αυτά τα προσωρινά αποτελέσματα, θα αρχίσω να εργάζομαι πάνω στο τεχνικό έγγραφο. Και να μπορέσουμε να μεταφραστεί το κείμενο, ελπίζω ότι μεταξύ κάπου γύρω στα 15 και 16 θα μπορέσουμε να σας μοιράσουμε και το τελικό κείμενο για να είμαστε σίγουροι ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα μπορέσει να το συζητήσει στις 29 και 30 Νοεμβρίου. Σημαντικέ ημερομηνίε αυτές για μα, λοιπόν. Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό έγγραφο πριν αρχίσουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Αυτό το χρονοδιάγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε στις 9 Δεκεμβρίου πάνω στο κείμενο, εδώ, και με το πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα θα μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε στην επόμενη συνοδομελία μετά αυτό το χρονοδιάγραμμα που προβλέπω. Έχουμε βέβαια ενδεχομένω προβλήματα με τη μετάφραση των κειμένων, αλλά ελπίζω να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Εκτός από τα τεχνικά αυτά θέματα, θέλω να προσθέσω ένα πράγμα. Οι απόψει μου παρουσιάζονται ξεκάθαρα στα δύο έγγραφα εργασία που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα. Το μόνο που θα ήθελα να πω εδώ όσον αφορά την έκθεση Κόμπολη. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε συναντηθεί με του εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών για το θέμα αυτό και ελπίζω να πάρουμε ένα κείμενο την επόμενη εβδομάδα. Για τρεις ε, εισηγητές δεν ήταν καλό αυτό. Η μόλις, είπε ότι θα μπορούσε, άλλοι εισηγητές δεν μπορούν. Αλλά εγώ προσβλέπω στον άγχο των το των να τα έγραφα στα χέρια μου. προς όφελος των άλλων μελών όμω που δεν έχουν παρακολουθήσει από στενά την έκθεση, θα πω ξεκάθαρα τι συμβαίνει και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η έκθεση είναι διαφορετική από τις άλλες εκθέσεις που έχουν ε, συζητηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Τα 5-6 έγγραφα που είχαμε στο Κοινοβούλιο με πολλές μας λεπτομέρειες για τους διάφορους ε, παράγοντες που οδηγούν στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. έχω να πω ότι αυτό το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ένα δυνάμει πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον των Ρώμα. Αυτό είναι το θέμα που μας ε, απασχολεί και πάνω σε αυτά η μελέτη θα μπορέσει να μας δώσει πολύ καλύτερα τις νομικές βάσεις που υπάρχουν και που μπορούμε να εξετάσουμε Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα πάνω στο οποίο ελπίζω να ακούσω τις απόψεις σας. Για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αποστείλουμε ένα πολύ α, ισχυρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας και πραγματικά ελπίζω όλοι οι βουλευτές να συμφωνήσουν. Είμαι λοιπόν ανοιχτή σε όποιες προτάσεις έχετε να κάνετε. Είμαι ανοιχτή για επιμέρους ε, συναντήσεις και εκτός από τους πιο συλληγητής ακόμα και την κοινωνία των πολιτών θα ήθελα να συναντήσω. Προσβλέπω λοιπόν σε αυτά και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Γερόκα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε πλέον τις μίας ευκαιριών να συζητήσουμε το θέμα αυτό διαμακρών. Και θα το ξανακάνουμε στις 26 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε τις προκατατικά αποτελέσματα της μελέτης. η οποία ξεκίνησε από την Κομισιόν και θα έχουμε κάποιες ευκαιρίες να επισέλθουμε στις σε αυτό το κείμενο. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτή τη στιγμή συζήτησή μας να εξετάσουμε το θέμα της παρουσίασης του εγγράφου εργασία και ακούσαμε από την εισηγήτρια όσα έχει να μας πει. Ίσως η Βελική Προεδρία, η Κομισιόν θέλει κάτι να πει πρωτού ανοίξουμε τη συζήτηση με τους βουλευτές που έχουν χτίσει το λόγο. Κομισιόν. Εάν όχι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Φίξτρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί που έχουμε επιτέλου ένα έγγραφο για τόσο σημαντικό αυτό ε, θέμα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση όπως το αποφάσισε η ΛΥΜΠΕ ήδη πέρσι. Είναι χρήσιμα τα έγγραφα εργασία γιατί μα δίνουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε καλύτερα αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά όμως δεν ασχολούνται παρά μόνο με τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα που με λυπεί εμένα και γενικά την ομάδα μου, την άλτε. Είναι παράδοξο για μένα ότι ενώ γίνονται απελάσεις, προετοιμάζονται κατάλογοι με εθνοτικά στοιχεία των πολιτών ε, δεν την εντύπωση ότι εξετάζουμε τα πιο σημαντικά θέματα εν ώψη αυτών. Προσπαθούμε νομίζω να θάψουμε τα κεφάλια μας στην άμμο σαν σορφοκάμιλη. Θα ήθελα να ζητήσω από την συγκεκριμένη να εξετάσει τα θέματα αυτά και να βοηθήσει έτσι τα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει πόσο νόμιμα είναι τα εκάστοτε εθνικά μέσα, πόσα αυτά τα χρησιμοποιούνται και ποιε είναι οι επιπτώσει του, τι γίνεται με τη στέγαση, τι γίνεται με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται με τι διακρίσει, με την απομάκρυνση από το υπόλοιπο τη κοινωνία. Τι μπορεί και πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιβιώσει ότι το θέμα της έκθεσης είναι η ένταξη στην κοινωνία των Ρώμα. Να μην έχουμε πια διακρίσεις για θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας η ομάδα Όλντε, μα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να εγκρίνει την έκθεση. Αλλά αυτή είναι περιττή κατά τη γνώμη μας αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κούντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα αναφερθώ σε δύο πτυχές της έκθεσης. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση αυτή γιατί την περιμένουμε πολλούς μήνες τώρα είναι σημαντικό να έχουμε κάτι επιτάπητος που μπορούμε να τροποποιήσουμε, να βελτιώσουμε κλπ. Και ελπίζω να έχουμε σύντομα μια συνάντηση με όλους τους κοιόδης συγητές. Έχω ε, προσφέρει διάφορες δυνατότητες συνάντησης στη Λίβια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι και η Επιτροπή Απασχόλησης θέλει να γνωμοδοτήσει και εγώ θα είμαι ε, στην Επιτροπή αυτή ή υπεύθυνη εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. θα μπορούμε από όλες τις πτυχές, το είπε και η Σεσίλια, να δούμε και την πτυχή της ασφάλειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας κλπ. Και καταρχήν θα πρέπει να εργαστούμε για το μέλλον και να φροντίσουμε να έχουμε κείμενα που είναι προς όφελος της ε, κοινότητας του Ρώμα. Μετά έχω να πω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι κάπως πολύ στενό. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστεί. Και έτσι η το προθεσμία της τροπολογίας θα πρέπει να είναι κάπως για τα μέσα Δεκεμβρίου και θα χρειαστούμε μετά και χρόνο να εξετάσουμε τροπολογίες, να προετοιμάσουμε συμβαστικές τροπολογίες. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να συζητήσουμε και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των Ρώμα. 25, 25 ε, Ιανουαρίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Δηλαδή αναβάλουμε κάπως το χρονοδιάγραμμα αυτά. Θα εξαρτηθεί και βέβαια από τις μεταφράσεις. Αλλά να ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και θα δούμε μετά πότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην ολομόλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλο. Συμφωνώ με την Τσεσίλια Μαξ. Um, on the issue of discrimination, which I see is very much missed. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που λείπουν από την έκθεση γιατί δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει η ενσωμάτωση των ατόμων αυτών. Υπάρχουν και έντονε διακρίσει κατά τον Ρώμα σε όλε τι κοινωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, να σταματήσουμε τι διακρίσει με οποιαδήποτε μέσα μπορούμε και δεν το βλέπω αυτό στο έγγραφο εργασία προ το παρόν. Επίση δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπίσει το θέμα φύλου στην τελική σα έκθεση. Και θα ήθελα επίση να συγκεντρώσω και προσοχή σα περισσότερο στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση και η ένταξη στην κοινωνία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεν είναι μόνο το τι κάνουν οι Ρώμα, αλλά και ότι πρέπει θα προσφέρουν οι μη Ρώμα, αν μπορώ να τι πω έτσι, κοινωνίες. Πώς θα αλλάξουν εκείνη τη συμπεριφορά τους, ο τρόπο με τον δρούν, τι θα προσφέρουν, πώ θα μπορούν να διευκολύνουμε την ε, ένταξη στη σχολεία των παιδιών Ρώμα. Χωρίς να σου λέμε ότι θα πρέπει να μείνετε τώρα εδώ και να μην κουνήσετε από αυτόν τον τόπο για τα επόμενα 7-10 χρόνια που θα στο σχολείο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια εμφιότητα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κλής. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Υποθέτω ότι στο έγγραφο της κυρίας Γιαρόκο χρησιμοποιείται πιο επίσημη γλώσσα από ότι στο κείμενο που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια. Είναι θετικό και πιστεύω επίσης θετικό ότι μιλάει και για το κόστος της μη ένταξης των Ρώμα. Το κείμενο αυτό πάντως θα κερδίσει σε αξιοπιστία εφόσον Μιλάμε και για την ευθύνη που μπορούν να πάρουν οι ίδιοι οι Ρώμα. Γιατί πάντα λέμε, κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος το Ρώμα, ενώ διάφοροι ειδικοί και στην Ολλανδία αλλά και στην Φλάνδρα έχουν πει ότι μέσα στους ίδιους τους Ρώμα Υπάρχουν θέματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει. Για παράδειγμα, η σχολική αποτυχία. Γιατί, γιατί τα παιδιά πηγαίνουν πολύ λίγο στο σχολείο, δεν πηγαίνουν αρκετά χρόνια στο σχολείο. Ή οφείλεται επίση στο ότι η... τα κορίτσια παντρεύονται πάρα πολύ μικρά στην ηλικία. Ή γιατί αναγκάζουν πολλοί γονεί τα παιδιά τους να πηγαίνουν και να ζητιανεύουν. Και μερικές φορές ανακατεύονται και σε εγκληματικέ δραστηριότητες. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να φροντίσουμε για αυτά τα θέματα να συζητήσουμε με τους Ρώμα έτσι ώστε να αναλάβουν και αυτή την ευθύνη. Να μην μιλάμε μόνο για δικαιώματα που έχουν οι Ρώμα αλλά και για υποχρεώσεις που έχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άνσιο. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να τελειώνουμε πια με την ολοκλήρωση των Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάτε ότι και αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που δημιούργησε τόση δυσαρέσκεια. Θεωρώ και δεν θέλω βέβαια να μπω σε λεπτομέρειες για το έγγραφο εργασία, πιστεύω έλεγα ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ για τις ειδικέ οικονομικές συνθήκες των χωρών όπου κατοικούν οι περισσότεροι Ρώμα. Όταν οι Ρώμα φεύγουν από αυτή τη χώρα, δεν είναι ότι τους αρέσει πια τόσο πολύ να πηγαίνουν να μένουν σε στρατόπεδα χωρίς συνθήκες υγιεινής και με αυτή τη χάλια κατάσταση. Προσπαθούν οι άνθρωποι να διαφύγουν από τη φτώχεια στη χώρα προέλευσης. Μιλήσατε και για το ποσοστό της εγκατάλειψης των σπουδών, που είναι πολύ ψηλό. Να σας δώσω όμως εγώ το αντίθετο αποτέλεσμα το ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών από τους Ρουμάνους μη Ρώμα είναι μεγαλύτερο από εκείνο το Ρώμα. Βέβαια όλα είναι πολύ πιο δύσκολα για τους Ρώμα από ότι για τους άλλους, ακόμη και για το θέμα της ε, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Στη Ρουμανία το σύστημα υγείας είναι κατεστραμμένο. 22 εκατομμύρια κάτοικοι δεν, ναι, δεν μπορούν να, να υποφεληθούν από ένα σύστημα υγείας, πόσο μάλλον η Ρώμα. Η κατάσταση δε της ανεργίας είναι χάλια. Λόγω της ανεργίας είναι αδύνατον η Ρώμα να βρουν οποιαδήποτε δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν φεύγουνε. Πρέπει λοιπόν εμείς να κοιτάξουμε ούτω ώστε η Ρώμα να μην είναι η φτωχή μεταξύ των φτωχών. Ο κ. Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας είναι μια πολύ καλή αρχή για τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Υπενθυμίζω και εγώ ότι το ζήτημα των Ρωμά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Αναφερόμαστε σε Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετική γλώσσα σε κάθε χώρα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικές συνήθειες, ήδη έθιμα, όλα αυτά κάνουν ακόμη πιο σύνθετη την ε, στη διαβούλευση που έχουμε να κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό καθ' όλη αυτή την περίοδο που έχουμε μπροστά μας να είμαστε νυφάλοι και να, μην, και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις εξάρσεις και να λειτουργούμε σε κλίμα συνένεσης. Και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο η κυρία Γιαρόκα συμβάλλει καθοριστικά. Εγώ πραγματικά την ευχαριστώ για όσα μέχρι σήμερα έχει κάνει και προκαταβολικά για αυτά που θα κάνει Ξέρουμε ότι κατάγεται από τους Ρωμά και παρόλα αυτά δεν υιοθετεί ένταση στις τοποθετήσεις της. Το αντίθετο κάθε φορά πολύ ισορροπημένα θέτει τα ζητήματα και πραγματικά αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Νομίζω κυρία Γιαρόκα ότι και εσείς σε αυτή την προσπάθεια έχετε την ευθύνη, τη σκέψη μας κάποιες φορές να την οδηγείτε προς τα σημεία που πρέπει να δίνουμε τη μεγαλύτερη προσοχή. Και ε, κλείνοντας μια ιδέα μόνο θα ήθελα να θέσω, το κουβεντιάσαμε αυτό και μια άλλη φορά. Ε, μήπως, επειδή υπάρχουν, συζητάμε για, την, ε, για το ότι δεν πρέπει να έχουμε διακρίσει, συζητάμε για τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν στι κοινότητε στο Ρωμά και θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα και πρότυπα για ενσωμάτωση, μήπως θα ήταν καλή ιδέα σε κάποια από τις συνεδριάσεις μας να προσκαλέσουμε και κάποιον που είναι Ρωμά και έχει διακριθεί και έχει προχωρήσει τη ζωή, αποτελεί πρότυπο ενσωμάτωσης και μέσα από ένα τέτοιο διάλογο να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε επιπρόσθετα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Κυρία Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Υπό το φως των γεγονότων των τελευταίων εβδομάδων και ημερών σε μια χώρα μέλος που γνωρίζω πολύ καλά, ε, βγήκε και κάτι καλό. Ότι μπορούμε να σμπρώξουμε λίγο τα πράγματα και να περάσουμε σε μια ψηλότερη, με μεγαλύτερη ταχύτητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΡΟΜ. Βέβαια η Ρώμα ποτέ δεν θα είναι, δεν θα είναι άμυρη παρεξηγήσεων και παρερμηνιών. Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε σε σαφείς προτάσεις ούτως ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παρερμηνίας αυτών των διατάξεων από οποιοδήποτε κράτος μέλος για τα θέματα ένταξης στο Ρώμα στα κράτη-μέλη. Υπέβαλα λοιπόν τροπολογίες αυτή την έκθεση, ούτω ώστε μερικά θέματα τα οποία απλώς θα επενήσεται η έκθεση να ενισχυθούν και να βοηθήσουν στο μέλλον να προχωρήσει η κατάσταση. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνετε, Λίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγισή σου, που είναι ευρεία. Για να βρούμε μία βάση για κοινή στρατηγική απέναντι στους Ρώμα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί οι τελευταίες εξελίξεις έδειξαν ότι η Ευρώπη τη χρειάζεται αυτή την κοινή στρατηγική. Δεν είναι θέμα της Ρουμανίας, δεν είναι θέμα της Σλοβακίας, δεν είναι θέμα της Ουγγαρίας ή των Ισπανών, Ρώμα κλπ. Είναι θέμα της Ευρώπης πώς θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι για να αποφύγουμε να βάλουμε τα πάντα στην έκθεση που θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο και σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Για να το αποφύγουμε αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στη στρατηγική, τι δηλαδή θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να κάνει για αυτήν την ομάδα Ευρωπαίων πολιτών και από την άλλη τι έχει να κάνει με την επιβολή του νόμου. Τι λέει ο νόμος στην Ευρώπη, είναι ανάγκη να τον χρησιμοποιούμε τον νόμο, να τον εφαρμόζουμε και στην περίπτωση των Ρώμα. Αλλά αυτά είναι δύο χωριστά, διακριτά θέματα. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μποσκούρτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν εκεί οι υπόλοιποι, αλλά έχω να προσθέσω μερικά και να υπογραμμίσω. Πρώτα απ' όλα, αυτό που μόλις είπε η κυρία Μπάουερ, ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τα δύο ζητήματα. Να δούμε τι είναι αυτό που έχει να κάνει με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για 12 εκατομμύρια ανθρώπου στο κάτω-κάτω που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φροντίσουμε και για την κοινωνική τους ένταξη. Είναι καλό λοιπόν η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που ξεκινάει μια γνωμοδότηση για αυτό το θέμα αυτό το οποίο δεν βρίσκω στο έγγραφο εργασίας. Και συχνά το έχουμε πει αυτό, είναι ποια είναι η εκπροσώπηση των Ρώμα. Άμα θέλει κανείς μια στρατηγική, καλό είναι η ίδια η ομάδα για την οποία γίνεται η στρατηγική αυτή να συμμετέχει. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά στην πράξη δεν γίνεται σχεδόν τίποτα από αυτού. Η Ρώμα είναι ένας εύκολος αποδιοπομπαίο τράγος όπως το έχουμε δει στην πράξη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε εφόσον θέλουμε μια στρατηγική να το συμπεριλάβουμε. Και τέλος, μην ξεχνάμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και με τις υποψήφιες προσένταξη χώρες για να αποφύγουμε προβλήματα είτε πρόκειται για τη Βοσνία, είτε για την Σερβία, να φροντίσουμε να δούμε πώς μπορούν και αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν στην εκπόνηση μιας στρατηγικής, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την πιο σωστή λύση, που θα είναι και διαρκείας. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, η συγκήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη, γιατί βλέπω ότι πέρασε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για μένα. Θα ακολουθήσω τις προτάσεις σας. Για να βεβαιωθούμε ε, πώς πρέπει να έχει έκθεση. Στόχος της έκθεσης και δικός μου στην έκθεση αυτή είναι να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική ευρωπαϊκή για τους Ρώμα. Το δεύτερο είναι τι πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική αυτή. Οπότε θέλω να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής αυτής να επικεντρωθούν σε αυτό. Να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την νομική πτυχή και την άλλη. Και στην αρχή αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία λέω ότι η εφαρμογή των οδηγιών που έχουμε σήμερα, η καλή εφαρμογή των οδηγιών που έχουμε σήμερα θα είχε οδηγήσει, θα οδηγήσει από εδώ και πέρα στο να μην έχουμε τέτοια ε, προβλήματα, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ με την στρατηγική αυτή είναι ένα μέσο ακριβώς γι' αυτό στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Θέλω όμως ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, προβλήματα συνενώσεις μερικές φορές, να έχουμε και τα κονδύλια που χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Τα πιο σημαντικά πέντε σημεία μου είναι νομική βάση, μια χαρτογράφηση της κρίσης που είναι δηλαδή, τι προγράμματα υπάρχουν, αλλαγές σε εδαφικό επίπεδο, να δούμε τι αλλάζει στην κατανομή και εκεί μπορούμε να ακούσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να φτιάξουμε αυτή τη χαρτογράφηση που σας έλεγα που βρίσκονται οι Ρώμα και πώς μετακινούνται. Και έπειτα θέλουμε και τους χάρτες αλλά και τα προγράμματα δράσης που τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρώμα. Εγώ δηλαδή θέλω να φροντίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το εύρος της έκθεσης λοιπόν είναι αυτό που σας είπα. Αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα. Το οικονομικό, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης πριν από λίγα χρόνια, οικονομολόγος που ήρθε και μίλησε εκεί και έχω συμπεριλάβει αυτά που είπε στην έκθεσή μου. Όπως και το θέμα των δύο φύλων. Είναι και αυτή μια διάσταση που μας φέρνει η Επιτροπή για τα Δικαιώματα ε, των Γυναικών και η Περιφερειακή Επιτροπή επίσης έχει να προσφέρει. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες επιτροπές που έχουν λόγο στην έκθεση αυτή. Υπάρχει μια άλλη πτυχή στην οποία αναφερθήκατε, πολλοί από εσά που είναι η υπευθυνότητα των ίδιων των Ρώμων. Τι, δηλαδή μπορούν εκείνοι να κάνουν, πώς μπορούν να συμμετέχουν Είδατε ότι θέλω μια έκθεση ισορροπημένη. Και ακόμα και αν έχουμε μια στρατηγική για τους Ρώμα, αυτό θα είναι 10%. Ένα 20% θα έρθει από τα κράτη-μέλη, ένα άλλο ποσοστό θα έρθει από τις τοπικές ε, αυτοδικήσεις και ένα 50% θα λέγω ότι θα έρθει από τους ίδιους τους Ρώμα. Πως εκείνοι θα ελέγξουν την εφαρμογή των προγραμμάτων και της στρατηγικής που προβλέπετε για τους ίδιους. Όντως, η νέα γενιά, κυρία Μποσκούρτ, πρέπει να συμπεριληφθεί για να πετύχει η στρατηγική μας. Όταν θα έχουμε το πλαίσιο που εγώ προτείνω, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν και άλλες εκθέσεις από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση να δώσει τη σωστή βοήθεια και ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο ώστε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Πολλά ζητήματα μένουν ανοιχτά δηλαδή. Πάντως με την έκθεση αυτή, αν μη τι άλλο, θα δείξουμε το δρόμο που πρέπει να πάρουμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε για να πετύχουμε. Να φροντίσουμε να συμπεριληφθούν όλες οι πλευρές. Αν πιστεύετε ότι η έκθεση πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να λέει περισσότερο τι πρέπει να κάνουν οι Ρώμα ή μη Ρώμα, εντάξει, τα κράτη-μέλη, οι πολιτικοί, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να τηρήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη. Είναι πολύπλευρο δηλαδή το θέμα και στην έκθεση αυτή πρέπει να φανεί ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από ότι μια καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζονται και άλλα. Και αυτό το επιπλέον που χρειάζεται είναι στα χέρια, στη γνώση εκείνων των πολιτικών που δουλεύουν στον οικισμό, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση. Μόνο τότε θα πετύχουμε, αν όλοι αυτοί συμπεριληφθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδέες που μου δώσατε και παρακαλώ βομβαρδίστε με με τις ιδέες σας μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Νταρόκαν. Ευχαριστούμε και όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Σας υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό στις 26 Οκτωβρίου θα μπει και πάλι στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, που είναι το σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη και που είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας 2003 κάθετο 109 στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Κλοντ Μωράε. για το θέμα αυτό, που είναι η επέκταση του καθεστώτος κατοίκων μακράς διαρκείας και στους πρόσφυγες. Ο κύριος Μωρέας θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα που είχε με τους σκιώδεις, της που είχε με τους σκιώδες συζητητές την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι ώστε να προετοιμαστεί ο πρώτος τριμερής διάλογος που θα λάβει χώρα στις 12 Οκτωβρίου. Αύριο δηλαδή. Κύριε Μωράης, έχετε το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είμαι γνώμων που έχουμε προχωρήσει. Θέλουμε η υποβελγικής προεδρίας να προχωρήσει το θέμα αυτό. Τα δύο στοιχεία κλειδί για τα οποία χρειάστηκε να συμφωνήσουμε οι σκιώδεις εισηγητές ήταν πρώτον κατά πόσο οι συγγενείς έχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ακολουθήσουν αυτούς οι οποίοι εκδιώχνονται. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια τροπολογία της Μαρίας Ανατοτσίβα που είναι εδώ, της Οσίλιας ε, Βάστρομ, της Αρτζεντίνη και μου του Ιδίου. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν πολλές φορές με την ενδοοικογενειακή βία. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ε, τα μέλη της οικογένειας να ακολουθούν κάποιον ο οποίος διώχνεται από τη χώρα. Δεύτερον, είχαμε δύο συμβαστικές τροπολογίες για την ε, έκδοση σε τρίτη χώρα, απέλαση μάλλον σε τρίτη χώρα, και αυτό γιατί αν δούμε πώς ερμηνεύεται το άρθρο 21, επιτρέπει απελάσεις να γίνονται σε τρίτες χώρες και εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός διαβούλευσης στο πρώτο και στο δεύτερο κράτος μέλος, για να δούμε τι λένε και αυτά. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, πιστεύω ότι εμείς προχωρήσαμε πολύ όσον αφορά τις διαφορές που είχαμε μεταξύ μας. Και πιστεύω ότι για τον τριμερή διάλογο είμαστε σε καλή θέση τώρα. Το Συμβούλιο είπαμε ότι θέλουμε να λύσει το θέμα σύντομα, να δούμε το θέμα του χρονοδιογράμματος όσον αφορά την αίτηση ασύλου. Σε μερικές χώρες καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία και διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Άρα λοιπόν ο υπολογισμός αυτός είναι ένα τελικό θέμα που μένει ακόμα να λύσουμε με το Συμβούλιο. Πάντως οι σκιώδεις είχαμε μια πολύ θετική εμπειρία. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους και την γραμματεία που βοήθησε πολύ και έτσι είμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τον αυριανό τριμερή διάλογο. Ευχαριστούμε κύριε Μωρές. Ξεκινάει η συζήτηση τώρα. Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ, κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ένα από του σκιώδες συζητητέ στο Dream Team του κ. Μουράς και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την γλίγορη τέλεση των εργασιών και το ότι συμπεριλάβα τι απόψει μας. Συμφωνώ ότι η αρχή του υπολογισμού του χρόνου θα πρέπει να ξεκινάει τη στιγμή που κάποιο για πρώτη φορά υποβάλλει την αίτηση. Επίση, θα ήθελα να ξελέω ότι ένα άτομο με ε, διεθνή προστασία ε, μπορεί να απελαθεί στην περίπτωση κατά την οποία ε, έχει, ανα, έχει πραγματοποιήσει κάποια κλιματική πράξη, αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να απελάσσονται και οι, τα μέλη της οικογένειας του. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και ελπίζω ότι θα τύχει επαρκούς εν, υποστήριξη αυτή η έκθεση και η τελική ψηφοφορία θα είναι επιτυχής και θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Συμβούλιο για την προσαρμογή τη έκθεση αυτή που θα ε, συμβάλλει ελπίζω στην επιτάχυνση διαδικασία και για τα άλλα θέματα της δέσμη. Και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής μέχρι το 2012. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στον τριμερή διάλογο αύριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκεώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ και θέλω να υποστηρίξω τον κύριο Μωράης, να τον ευχαριστήσω για τη επικοδομητική του αντιμετώπιση. Αυτό μας βοήθησε και την προηγούμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε ιδιαίτερα ισορροπημένες ε, αποφάσεις και συμβιβασμούς. Δύο συμβιβασμούς βρήκαμε. Για το θέμα της ε, ε, απέλασης των μελών οικογενείας είναι πολύ σημαντικό η εισδοχή, η επανεισδοχή των μελών της οικογένειας στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης να γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο ή με τους εθνικούς νόμους. Καταφέραμε να βρούμε όμως συμβιβασμό σε αυτό. Τώρα, για την απέλαση προς τρίτη χώρα, ο συμβιβασμός που βρήκαμε είναι επίσης πολύ ικανοποιητικός. Είναι, πρόκειται για τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών για να δούνε αν θα ε, υπάρχει ρίσκο δίωξης του απελαυνόμενου στην τρίτη χώρα. Και αυτό βάσει της οδηγίας ε, του 2000 Τέσσερα. Πιστεύω ότι αν καταφέρουν να συμφωνήσουν και τα τρία θεσμικά όργανα γύρω από αυτό το ντοσιέ, πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος για το πακέτο του ασύλου. Ευχαριστώ κυρία Νέλτσεβα. Εγώ δεν βλέπω κανέναν άλλο συνάδελφο να θέλει να μιλήσει. Βλέπω, βλέπω ικανοποίηση για το πώς έχει προχωρήσει ο Τρίλογος. Είναι ευχαριστημένοι όλοι και όλες. Σας ευχαριστώ. Να πάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο 6. 8. 8. Ελάχιστε απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώ των υπηκών τρίτων χωρών ή των απατρίδων ατόμων ω δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο τη have προστασία. Ε, η, συγγήτρια είναι η κυρία Τζιν Λάμπερτ που θα μας κάνει την παρουσίαση ενός σχεδίου έκθεσης για τροπή στις οδηγίες αυτής που είναι ένα από τα κύρια τμήματα της λεγόμενης δέσμιας σύλλου Θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και μετά θα ακούσουμε και την Επιτροπή ή την Προεδρία αν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, αλλιώς θα συζητήσουμε μεταξύ μας. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα θυμούνται οι βουλευτέ ότι οι περασμένη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα εξετάσαμε σε ένα έγγραφο εργασία πάνω στο θέμα αυτό που παρουσίαζεται τα κύρια συστατικά της οδηγίας αυτής. Ε, και επίσης εμείς δεν εξετάζουμε γενική προς οδηγίας, αλλά ορισμένα μεμονωμένα σημεία της, το ένα τους λόγους προστασίας των ε, εκείνων που ε, θεωρούνται ότι είναι ε, πρόσφυγες και εκείνοι που έχουν μια συμπληρωματική προστασία. Και ένα από τα κύρια θέματα που έχει πραγματοποιήσει η Κομισιόν εδώ είναι να συνενώσει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο προστασίας για τα οποία δεν ε, προτείνω και πολύ συγκεκριμένε τροπολογίε, γιατί πιστεύω ότι είναι ευθυγραμμισμένα με αυτό που θέλουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και που πραγματοποιούν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Δεχόμαστε λοιπόν εδώ τι προτάσει τη Κομισιόν, ίσω κάποιοι βουλευτέ να έχουν διαφορετικέ απόψει. Ε, έχω υποβάλει πολύ λίγες τροπολογίες. Η μία λύπη, ίσως το είδατε αυτό, υπήρχε μια αναφορά που υπάρχει ε, στην θεολογική σκέψη χωρίς να έχω υποφέρει συγκεκριμένη τροπολογία ακόμα. Ορισμένοι μου έκαναν την παρουσίαση και σας ευχαριστώ Όσο το διαβάσετε το κείμενο τόσο προσεκτικά που να μπορείτε να μου κάνετε την παρατήρηση αυτή. Αυτό που αναφέρεται στη μεθολογική έκθεση είναι μια μικρή σειρά τροπολογιών που αφορούν το θέμα του φύλου και σε αυτό το σφύλου όσον αφορά όταν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα πρόκειται για το άρθρο 29 και 11 δέλτα. Και επίση υπάρχει εδώ μία πρόταση που δείχνει μικρή αλλαγή. Δηλαδή αντί για ένα και συμπληκτικό υπάρχει ένα είτε διαζευτικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες διατάξεις που αφορούν κοινωνικές ομάδες με κοινά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο, το δεύτερο σημείο είναι ή είτε θεωρούν ότι είναι διαφορετικά από την ε, κοινωνία στην οποία ζουν. Δηλαδή δεν είναι συλλεκτικά, συλλεκτική λόγη αυτοί, είναι εναλλακτικοί. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ε, τροπολογία στο 10 ΔΕΛΤΑ. Υπάρχουν και άλλες μικρές τροπολογίες για διάφορα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του παιδιού. Υπάρχει ένα βασικό θέμα για τη συνέχιση της ενίσχυση των παιδιών. Αυτό τέλος πάντων δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά εκεί που στην Ευρωπαϊκή Σκέψη 17 η Κομισιόν προτείνει πιο έντονη διατύπωση για τα δικαιώματα των παιδιών, σύμφωνα και με τις διεθνείς συμβάσεις, εγώ προτείνω μια τροπολογία που λέει ποια θα πρέπει να είναι τα στοιχεία αυτά. Και προτείνω προτείνεται και ένα νέο άρθρο 2.1 που σχετίζεται με αυτή την ιδεολογική σκέψη 17. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που αφορούν τους ανήλικους, το άρθρο, η τροπολογία 10 για το άρθρο 2 δέλτα. Όπου αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους. Άλλο θέμα που ευθύγει είναι εκείνο που αφορά το άρθρο 7 και τις δράσεις προστασίας. Και όπως λέω στην εκτελική ε, έκθεση υπάρχουν πολύ έννοιες απόψεις εδώ από την UNHR, από, την... από άλλους τέλος πάντων ότι οι πράξεις προστασίας θα πρέπει να προέρχονται ε, μόνο από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα των φορέων προστασίας. Γιατί οι κυβερνήσεις διαφέρουν σε απόψεις τους. Εγώ προσπαθώ να έχω μία κάπως σχετιζόμενη τροπολογία για το άρθρο 7. Και αναφέρομαι εδώ στις τροπολογίες 6 και 7 που καθιστούν πιο αυστηρούς τους, τους όρους ε, ικανοτήτων εκείνων που ε, μπορούν να προσφέρουν την προστασία αυτή. Όχι μόνο από πλευράς, αλλά γιατί θα πρέπει να μπορούν να θεωρηθούν υπόλογοι και υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Ίσως θα μπορέσουμε να έχουμε μια διαφορετική διατύπωση του θέματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άρθρο 8 που αφορά την εγχώρια προστασία, το να κινείται κανένας στο εσωτερικό της χώρας, η πρώτη Κομισιόν προσθέτει θέματα αποτελεσματικής και μόνιμης προστασίας. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει αυτή η δοκιμασία που είχαμε στο παρελθόν. Αυτές είναι οι μόνες τροπολογίες που προτείνω αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα όρια του τι μπορούμε ή και δεν μπορούμε να πετύχουμε. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν άλλες τροπολογίες. Αυτά είναι όμως τα πιο σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λαμπέρτ. Αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο προωθεί η Επιτροπή για να υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν στις χώρες μέλη για το άσυλο και προκειμένου να υπάρξει ένα ενίο καθεστώς προστασίας. Οπότε είναι αναγκαίο το διάβημα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη όσον αφορά το άσυλο και τοποθετούνται διαφορετικά. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτό το κείμενο, αυτή η νέα οδηγία. Πάνω απ' όλα, πρέπει να δούμε στο καθεστώς των προσφύγων και της διεθνούς προστασίας να φροντίσουμε να υπάρξουν περισσότερα ωφέλη και ίδια δικαιώματα για τους ανθρώπους που ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βήμα που έχει γίνει με τις τροπολογίες της κυρίας Λάμπερτ. Θα ακούσουμε φυσικά ξανά και ξανά για αυτό το θέμα στο μέλλον. Όπως το θέμα των ε, ε, φυλάκων προστασίας κλπ. Η συνεισφορά της κυρίας Λάμπερτ, έστω και αν είναι ελάχιστη, είναι καλά τεκμηριωμένη. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε αυτές τις θέσεις. Τώρα, αν μπούμε στο θέμα του ασύλου, το θέμα του ασύλου είναι πολύπλοκο και οι διατάξεις. Επίσης το θέμα της ισόρευσης προσφυγών είναι πολύπλοκα αλλά και οι καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών είναι διαφορετικές ε, μεταξύ τους. Όλοι δεν έχουν τα ίδια σύνορα με καλές χώρες. Και κάθε χώρα έχει τις παραδόσεις της που είναι προσαρμοσμένες και με τη γεωγραφική τους κατάσταση. Αλλά οι χώρες που τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν χώρες υποδοχής για τους ετούντες ασύλου έχουν κλείσει αλλά πρέπει να δούμε γιατί και ίσως οι όλοι οι λόγοι δεν αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λάμπερτ για την πολύ καλή και ισορροπημένη δουλειά που έχει κάνει. Ε, ο εισηγητή τη ομάδα μα, ο κύριο Χολμάιερ, δεν είναι σήμερα μαζί μα. Για λογαριασμό όμω τη ομάδα μα, θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο, αν είναι εφικτό, να έχουμε κάποια παράταση σε ό,τι αφορά την κατάθεση τροπολογιών την, ε, ε, σας λέω μόνο το πρόβλημα που έχουμε στη δική μας ομάδα. Αύριο οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων θα βρεθούμε στην Πορτογαλία γιατί έχουμε ε, τα, τα study days εκεί, η δική μας ομάδα και επιστρέφουμε την Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το Στρασβούργο και γι' αυτό παράκληση θερμή για λογαριασμό της δικής μας ομάδας αν μπορούμε να έχουμε κάποιες περισσότερες ημέρες για να μπορέσουμε να εργαστούμε και να συνεισφέρουμε κι εμείς όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Thank you. Άλλα σχόλια, άλλες προτάσεις. Κανένας άλλος, ε, κομισιόν, προεδρείο, ε, ε, συμβούλιο, συγγνώμη. Ο κύριος εκ, με... εκ μέρους του Έλκα ο κύριος Παπα-Νικολάου ζήτησε. Συμφωνείτε με αυτό που ζήτησε κυρία Λάμπρεχτ για αναβολή των προθεσμιών. Δεν έχω αντίρρηση, λέει κυρία Λάμπερτ. Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν. Οπότε θα το ξαναδούμε με την γραμματεία για τις προθεσμίες και θα φροντίσουμε να τις προσαρμόσουμε. Για να ανακουφιστεί όποια πολιτική ομάδα θέλει. Θα τις ξαναδούμε λοιπόν τις προθεσμίες. Ωραία, σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Από ό,τι βλέπω και άλλες πολιτικές ομάδες θα συμφωνήσουν. Τουλάχιστον δεν θα αντιτεθούν στο αίτημα αυτό. Οπότε θα συμφωνήσουμε και θα δούμε εδώ με την γραμματεία πώς θα ορίσουμε τη νέα προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Σύμφωνοι. Καλώς. We thank you again. No further σας ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζουμε και περνάμε. Στο σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη, που είναι η πρωτοβουλία πολιτών. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σημείο 9, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Πρωτοβουλία πολιτών. Θέμα ουσίας που έχει να κάνει με τις συνταγματικές εξελίξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εδώ το σχέδιο γνωμοδότησης που ετοιμάζει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Και η Επιτροπή Αναφορών συμμετέχει βάσει του κανονισμού, βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού. Πρωτοβουλία πολιτών λοιπόν. Είναι μια σημαντική καινοτομία που έχουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η οποία επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία και στη δημοκρατική συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το θέμα αυτό της πρωτοβουλίας πολιτών που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για το πώς δηλαδή μια πρωτοβουλία πολιτών ε, μπορεί να προχωρήσει και να καταλήξει ένα αποτέλεσμα. Έχουμε δύο συνεισηγητές για την γνωμοδότηση αυτή. Έχουμε τη συνάδελφο Κίνκα Γκάντς και την κυρία Σεσίλια Βίλκστρομ. Θα μας παρουσιάσουν σήμερα την γνωμοδότηση εδώ στην Επιτροπή μας, Τι ΛΥΠΕ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στη συζητήτριες και μετά όποιος άλλος θέλει να συμμετάσχει, Ευχαριστώ να του δώσω το λόγο για να πει ό,τι έχει να πει. Τώρα, επειδή ο χρόνος προχωράει, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ήδη μια προθεσμία για αύριο, 12 Οκτωβρίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Αύριο, 12 Οκτωβρίου, στι 12 το μεσημέρι. Σύμφωνοι? Οπότε, η κυρία Βίλκστρομ να ξεκινήσει ή η κυρία Γκόντς, ποια από τις δύο πρώτα. Η κυρία Γκόντς πρώτα. Έτσι συμφωνήσαμε με τη Σεσίλια, ότι εγώ θα ξεκινήσω και μετά η Σεσίλια. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι η πιο σημαντική πτυχή της συνθήκης της Λισαβόνας. ενισχύει τη συμμετοχική δημοκρατία. Έχουμε κάποιες προτάσεις για τροποποίηση της πρότασης. Η βασική μας ανησυχία ήταν η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών να είναι όσο γίνεται πιο φιλική προς το χρήστη. Ξέροντας βέβαια ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές που να στηρίζουν μια τροπολογία. Οπότε οι βασικές μας προτάσεις είναι οι εξής. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη ηλικία για να μπορέσει κανείς να υπογράψει για μια πρωτοβουλία, να είναι τα 16. Ξέρουμε ότι η αρχική πρόταση ευθυγραμμιζόταν με την ελάχιστη ηλικία που έχει ένας ψηφοφόρος στην, ε, στις διάφορες χώρες. Όμως σε κάποιες χώρες μπορεί κανείς να ψηφίσει από τα 16, αλλού από τα 18, αλλού και σε μεγαλύτερη ακόμα ηλικία. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια ενιαία ελάχιστη ηλικία και προτείνουμε τα 16. Ένα από τα επιχειρήματά μας είναι ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται για μια διαδικασία λήψης απόφασης, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ένας πολίτης και στην οποία θα δώσει σάρκα και ωστά ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν εμείς να δώσουμε στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες για να συμμετέχουν στον ε, ευρωπαϊκό βίο. Ένα άλλο θέμα τώρα, μια άλλη πρότασή μας, είναι πώς συλλέγονται οι υπογραφές. Η αρχική πρόταση λέει το 1 τρίτο των χωρών μελών. Η εισοδίκη της Λισαβόνας λέει ένα μεγάλο μέρος των χωρών μελών. Πόσα είναι αυτά. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Εμείς Πιστεύουμε ότι το 1 τέταρτο των χωρών μελών φτάνει για να έχουμε συμμετοχή πολλών χωρών. Μια άλλη πρόταση έχει να κάνει για τις προθεσμίες. Μέσα σε τι χρονικό διάστημα πρέπει να μαζευτεί το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είναι όπως προτείνουμε εμείς τα τέσσερα χρόνια. Αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, οι οργανωτές λοιπόν της πρωτοβουλίας, εφόσον δεν στηρίζεται από λόμπις, από οργανώσεις κτλ. και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και τέτοιες πρωτοβουλίες, τα τέσσερα χρόνια που προτείνουμε εμείς δεν είναι και τόσο πολλά για να συγκεντρωθούν οι υπογραφές αυτές. Είναι ένα επίμαχο θέμα τώρα το πότε γίνεται παραδεκτή μια πρωτοβουλία. Εμείς λέμε ότι από 5.000 υπογραφές θα έπρεπε να είναι παραδεκτή μια πρωτοβουλία. Ακόμα και από μία χώρα μέλος γιατί οι πρωτοβουλίες για να μεταφραστούν, αν δεν έχει γίνει ακόμα ο έλεγχος ώστε να είναι παραδεχτές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε και μετάφραση και όλα. Εφόσον έχει κριθεί παραδεχτή μια πρωτοβουλία, τότε ναι, να μεταφράζεται και να συλλέγονται μετά οι υπόλοιπε υπογραφές. Πιστεύω ότι σε έξι μήνες μπορούν να έχουν συγκεντρωθεί χίλιες υπογραφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά να ελέγχει το παραδεκτό ή όχι της πρωτοβουλίας. Μια άλλη μικρή αλλαγή που θέλουμε εμείς είναι αυτό που αναφέρεται ε, ότι όταν μια πρωτοβουλία αντιβαίνει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε να μην κρίνεται παραδεκτή. Τώρα, θα ζητούσα από τη Σεσίλια να συνεχίσει για την συλλογή online, την επιγραμματική συγκέντρωση υπογραφών. Ευχαριστώ πολύ. Cecilia would continue with, with the data collection. Uh, Thank you, Mrs. Gons. Now we hear from our co Ευχαριστούμε. Η συνεισηγήτρια τώρα, η Σεσίλια Βίλκστρομ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπογράμμισα ποια είναι τα κύρια σημεία και άλλη φορά και τα είπε και συνάδελφος, αλλά θέλω να αποφελθώ από την ευκαιρία αυτή για να υπενθυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν κοινή γνώμη είχε εκφραστεί αρνητικά στα κράτη-μέλη μας για τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι πολιτικοί πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν σαν επιχείρημα την πρωτοβουλία πολιτών για να τους ενθαρρύνουν, να τους πούν δηλαδή ότι κοιτάξτε και εσείς θα έχετε ε, περισσότερο, περισσότερη δύναμη, θα έχετε μεγαλύτερο λόγο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ε, λοιπόν, τώρα μην καταστρέψουμε αυτή την ευκαιρία, μην γίνει καινή λόγου η υπόσχεση που δώσαμε για την πρωτοβουλία πολιτών, αντίθετα να τη χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να υψώνουν τη φωνή τους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, η, και, και εγώ θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χάρηκα πάρα πολύ που συνεργάστηκα μαζί της και ευχαριστώ πολύ και τις άλλες πολιτικές ομάδες που μας στήριξαν, ακόμα και αν σε κάποια ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, διαφωνούμε. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που έχουμε τη συζήτηση αυτή και που μου δίνετε ευκαιρία να σας ακούσω όλους. Και τελικά προφανώς θα τροποποιήσουμε τη γνωμοδότησή μας σύμφωνα με τις επιθυμίες ε, των συναδέλφων εδώ. Τώρα για, το, για την κεντρική ιστοσελίδα. Είμαστε πολύ δημιουργικοί όταν ξεκινήσαμε είπαμε ότι είναι ένας τρόπος με διαφάνεια οι πολίτες να μπορούν να κοιτάνε μια κεντρική στο σελίδα και να μπορούν εκεί να ενημερώνονται για όλες τις πρωτοβουλίες που συζητιούνται και για όλες τις πρωτοβουλίες για τις οποίες μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους, δηλαδή δίνοντας το όνομά τους, τα στοιχεία τους και ότι έτσι θα μπορούν να παρακολουθήσουν και όλη τη διαδικασία. Βέβαια, επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι πάντα μπροστά στον υπολογιστή τους και online, θα έπρεπε να επιτρέπουμε και την συλλογή υπογραφών σε χαρτί. Και τα δύο. Η συζήτηση τώρα είναι ποιος θα φροντίζει για την ιστοσελίδα αυτός, ποιος θα τη συντηρεί. Θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να είναι η Επιτροπή Αναφορών, Ποιο, Όποιος και να είναι, θα πρέπει να είναι μια κεντρική ιστοσελίδα, όπου οι άνθρωποι με διαφάνεια να μπορούν να δουν πόσε υπογραφές έχουμε σήμερα, πόσε θα έχουμε μετά από ένα μήνα, για κάποια πρωτοβουλία που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Αν έχετε ερωτήσεις, να μας τις πείτε. Και θα προχωρήσουμε στη σύνταξη της γνωμοδότησής μας αυτής ανάλογα με τις δικές σας επιθυμίες και προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχω εδώ πέρα ένα κατάλογο με ποιους θέλουν το λόγο. Πρώτο όμως, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει κάτι να μας πει. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τεντρέιρο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κάποια σχόλια. Θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία σημεία που είναι τα πιο επίμαχα. Ξεκινάω με την ιστοσελίδα. Φυσικά και θα υπάρχει ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα τη διαχειριζόμαστε εμείς. Και αυτή η ιστοσελίδα θα είναι και το Μητρό όπου συλλέγονται οι υπογραφές. Οπότε μπορεί κανείς έτσι να παρακολουθήσει πόσες υπογραφές υπάρχουν και σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ξέρουν οι άνθρωποι μέσω της ιστοσελίδας, ότι αξιολογεί την μία ή την άλλη πρωτοβουλία ή έχουν ήδη συλλεχθεί υπογραφές κτλ. Δεν πιστεύουμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των υπογραφών. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για μας η συλλογή υπογραφών είναι κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι οργανωτές φυσικά και με κάποια ιστοσελίδα και σε χαρτί, αλλά τότε πρέπει να φτιάξουν τη δικιά τους ιστοσελίδα. Για να τους βοηθήσει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει ένα λογισμικό το οποίο θα είναι open source, ανοιχτής πηγής, έτσι ώστε να μπορούν να το κατεβάζουν και να το χρησιμοποιούν για να συλλέγουν υπογραφές, να συγκεντρώνουν υπογραφές. Αλλά δεν θα είναι η Επιτροπή που θα κάνει τη συλλογή, ούτε που θα διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της ε, συλλογής υπογραφών. Τώρα για τον αριθμό, 5.000 υπογραφές. Εμείς καταλάβαμε ότι υπήρχε μεγάλη αντίσταση στην ιδέα αυτή. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που θα αποφύγουν να υπάρχει έστω και κάποιος αριθμός υπογραφών. Προσπαθούμε με τους εισηγητές να δουλέψουμε πάνω σε μια λύση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να κάνει από την αρχή της ε, πρότασης να επαληθεύει ό,τι πρέπει να επαληθεύσει, να φτιάξουμε δηλαδή ένα κατάλογο με τα κριτήρια που θέλουμε να εφαρμόζουμε, ώστε να μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινάμε. Τώρα 48 μήνες αυτή είναι μια νέα ιδέα, τα τέσσερα χρόνια δηλαδή. Είχαμε πει 12 μήνες, μετά είχαμε πει 18 μήνες. Πρώτη φορά ακούμε για 48 μήνες προθεσμία προκειμένου να συγκεντρωθούν οι υπογραφές που χρειάζονται. Πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό και κατά πόσο είναι επιθυμητό να αφήνουμε πρωτοβουλίες έτσι να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο θέλαμε μικρότερο χρονικό διάστημα. Πόσο πιο σύντομο δεν ξέρω, το συζητάμε. Αλλά 48 μήνες μας φαίνεται μεγάλο διάστημα. Κάτι άλλο που έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε πει τις απόψεις μας είναι το εξής. Το 1 τρίτο κρατών μελών, λέμε εμείς, πρέπει να συμμετέχει στην αρχική συλλογή υπογραφών. Συζητήθηκε και στο Συμβούλιο το Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι σωστό, όπως επίσης και το θέμα της ηλικία από την οποία μπορεί κάποιος να προτείνει την υπογραφή του για μια πρωτοβουλία. Να είναι δηλαδή η ηλικία από την οποία ψηφίζει γενικά ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά όμως τα συζητάμε με τους συζητητές και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τελέιρο, η συζήτηση τώρα. Η κυρία Εντερφέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις προτάσεις των εισηγητών, γιατί προσπαθούν να μειώσουν το κατόφλι για την συμμετοχή στην πρωτοβουλία των πολιτών. Αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη για την πρωτοβουλία αυτών των πολιτών, δημιουργούμε τεράστιε προεδοδοκίε. Πολλοί έχουν εντύπωση ότι αυτό πρόκειται για ένα δημοψήφισμα όπου οι πολίτε παίρνουν την απόφαση. Και ο που γοητεύσει είναι τεράστιο. Γιατί η επιτυχία μια πρωτοβουλία πολιτών δεν εξαρτάται τόσο πολύ από το πώ οργανωθεί η συλλογή των υπογραφών, αλλά από την αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ειλικρινά, βλέποντα Πώς ανταποκρίνεται η Κομισιόν σε ένα άλλο δημοκρατικό μέσο, ε, κοινοβουλευτικές δηλαδή, δεν έχω πλήρη εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και ότι όπως οποιοδήποτε άλλο εκτελεστικό σώμα και δημόσια διοίκηση, η Κομισιόν ε, απαντά στις ε, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με ένα καταπληκτικό τρόπο, καλλιτεχνικό θα έλεγα, με το να μην δίνει απαντήσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, εδώ θα δημιουργήσουμε επίσης προσδοκίες και θα υπάρχει τεράστια απογοήτευση των πολιτών. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και αναφορές στο παρελθόν, γιατί εδώ αυτό είναι μια αναφορά. Παραδείγματο χάρη οι νέοι που ε, υποβάλλουν ερωτήσει στο δίκαιο είναι πάρα πολύ ικανοί. Υπήρχε μια αναφορά που ε, ξεκίνησε από την κυρία μας, ε, ένα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ε, αναφορά που είχε τον τίτλο «Μία έδρα», μία έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συνέλεξε ένα εκατομμύριο και πάνω οι υπογραφές και η οποία δεν αποδώσει τίποτα. Αντί λοιπόν να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες για τη συλλογή των ε, υπογραφών, θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε σίγουροι θα λάβει σοβαρά υπόψη η Κομισιόν της, ε, την πρόταση αυτή. Για να δούμε η κυρία Κορατσαπέλη τώρα. Ευχαριστώ. Ε, Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία με την Κίγκα, με τη Σεσίλια και με τους ηγητές από τις άλλες ομάδες. Πλησιάσαμε πολύ σε αυτό που είπε ε, συνάδελφος εδώ, ότι το θέμα είναι να μην δημιουργούμε προσδοτικές και να οδηγούσουμε τους πολίτες σε απογοήτευση. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν, αλλά θέμα πώς θα χωρίσουμε τους κανόνες και πώς θα προωθήσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών και θα την καταστήσουμε σε μια πραγματική δυνατότητα άμεσης και ανοιχτής δημοκρατίας. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια φιλική προς το χρήστη διαδικασία, μη γραφειοκρατική, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θα ήταν καλό ως η Κομισιόν να αναλάβει, να οργανώσει μια ε, εκστρατεία ενημέρωσης ίσως. Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνη η Κομισιόν για τη συλλογή των υπογραφών. Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια διαφορά μεταξύ το να είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των ε, υπογραφών μια ομάδα πολιτών και η Κομισιόν να είναι υπεύθυνη μόνο για την καταγραφή κλπ. Γιατί Εάν η Κομισιόν συνέλεγε τις, πληροφο... τις υπογραφές θα ήταν μια πρωτοβουλία της Κομισιόν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κάποιοι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι οι οργανωτές και η οικονομική ενίσχυση και η διαφάνεια το ποια χρηματοδότηση θα δοθεί από ποιον, πότε, σε τι ύψος κλπ. είναι πάρα πολύ σημαντική για να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δεχτούμε κάποιον από μια τρίτη χώρα, ας πούμε, να πληρώνει τεράστια ποσά για marketing κάποιου προϊόντος. Πρέπει να υπάρχει εδώ απόλυτη διαφάνεια. Δεν θεωρώ ότι η εκμεγμένη πολιτική που είναι μέλη της ε, ε, προσωπικής ε, δημοκρατίας θα πρέπει να μπορούν να είναι εκείνοι που ξεκινούν τη διαδικασία αυτή. Γιατί εμείς έχουμε δυνατότητα να ξεκινήσουμε κάποια νομοσχέδια ήδη και άλλο η δημοκρατία και άλλο η άμεση δημοκρατία. Συμφωνώ με την Κίνκα και τη Σεσίλια ότι δεν λέμε ένα τέταρτο κρατόμελό, θα μπορούσαμε να πούμε ένα τρίτο. Για την ελάχιστη ηλικία διαφωνώ. Γιατί πραγματικά δεν θα ήταν ρεαλιστικό Ε, να υποχρεώσουμε όλη την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστρίας. Ούτε μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ελέγξουν τις υπογραφές βασιζόμενοι σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει, γιατί το μόνο σύστημα που υπάρχει ε, είναι το σύστημα των υποκριτικών καταλόγων. Και αλλιώ είναι και τυχαίο, γιατί να πούμε 15 και να πούμε 16, να πούμε 17 και μισό, να μην πούμε κάποια άλλη ηλικία. Ένα έτος όπως λέει η Κομισιόν είναι καλό, τέσσερα χρόνια δεν θα ήταν καλό γιατί θα χάνα την ορμή τους οι πολίτες. Και συμφωνώ με την πρόταση των ζητών Αύκα και Πέτρη να μειώσουμε ε, τα διάφορα βήματα για την καταγραφή και την, ε, το αποδεκτό κλπ. Γιατί αλλιώς θα ε, μπλεχθούμε με 5.000, 10.000, 100.000 υπογραφές. Και δύο ακόμα πράγματα με την άδειά σα, ε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι Ιταλίδα, αλλά κατοικώ στην Σουηδία. Ε, ξεχάστε ότι είμαι εκλεγμένο μέλο του κοινοβουλίου. Αν δεν ήμουν, α πούμε, ήμουν μια απλή πολίτη. Τι θα μέτραγε, η ηθαγένειά μου, η υπηκότητά μου ή που κατοικώ και τι γίνεται με Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν σε μια τρίτη χώρα, στην Αργεντινή, στη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει νομίζω να συμπεριλάβουμε και τα δύο αυτά στοιχεία. Και την υπηκότητα και τον τόπο διαμονής. Και επίση θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την απογοήτευση, την απώλεια των προσδιοκών κλπ. Διότι εάν έχουμε συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές και η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να πει δεν ενδιαφέρομαι να προωθήσω το θέμα. Τι θα κάνουμε. Υπάρχουν διάφορε ειδικέ προτάσει και θα πρέπει να τι συμπεριλάβουμε στην γνωμοδότησή μα. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Καρατσαμπίλτ. Λέει ο κύριος Κλάς ε, που είναι σκιώδης εδώ θα θέλει να μας πει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες εδώ που θέλουν να χαμηλώσουν το όριο. Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει. Βλέπετε, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί μέρος της ηθίκης της Λισαβόνας, αλλά που είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει απόλυτα. Έχουν την εντύπωση οι άνθρωποι ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του δημοκρατικού ελλείμματος. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει και εμείς με τα όρια που βάζουμε να δυσκολεύουμε την πρωτοβουλία. Οι διάφορες οργανώσεις, τα συνδικάτα κτλ. πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν εύκολα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, η προθεσμία μέσα στην οποία συγκεντρώνονται υπογραφέ. Συμφωνώ να είναι πιο μεγάλη. Είμαι όμω κατά τη τροπολογία αριθμό 3 των εισηγητών, εισηγητριών. Για το παραδεκτό. Βάση των ε, ευρωπαϊκών αξιών. Αν κάτι παραβαίνει, δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αρχές, τότε να μην γίνεται παραδεκτή. Εμείς όμως που νομοθετούμε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί τι σημαίνει αυτό. Συγκαλυμμένα λέει η τροπολογία μιλάει για καταχώρηση προτάσεων κατάφορα ή συγκαλυμμένα αντίθετον με τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει. Ανοίγουμε έτσι την πόρτα σε αυθαίρετες ε, αποφάσεις. Τι θα πει συγκαλυμμένες αντιθέσεις. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Γιατί τι θα γίνει σε όλες αυτές τις επίμαχες περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λέει ότι κάτι συγκαλυμμένα είναι αντίθετο στις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι όχι. Εμείς που είμαστε νομοθέτες πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε κριτήρια τα οποία είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα και όχι ασαφή. Και έχω και άλλη μία παρατήρηση σχετικά με τον αριθμό ταυτότητας των ατόμων που υπογράφουν. Στο κείμενο της Επιτροπής λέει ότι όταν υπογράφεται μια πρωτοβουλία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, την ηλικία, ε, τον τόπο κατοικίας και έναν αριθμό ταυτότητας, διαβατηρίου, κοινωνικής ασφάλισης, κάτι. Αυτά τα πράγματα τρομάζουν τους πολίτες και θα τους αποτρέπουν από το να υπογράψουν μια πρωτοβουλία. Εμείς θέλουμε να συγκεντρώνονται υπογραφές και όχι να υποχρώνουμε τους ανθρώπους να δίνουν πολλά περίπλοκα στοιχεία, ένας ο κόσμος δεν ξέρει καν ποιος είναι ο ρυθμός της κοινωνικής του ασφάλισης. Μην δυσκολεύουμε λοιπόν τα πράγματα, μην ανεβάζουμε τον πύχη και αποτρέπουμε τους πολίτες από το να δίνουν την υπογραφή τους για τις πρωτοβουλίες αυτές πολιτών. Δεν θα πρέπει λοιπόν με το κριτήριο αυτό να αποτρέπουμε τον κόσμο από τον υπογράφη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Αλβάρο τώρα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τις ζυγητρίες. Το έχετε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και μάλιστα μια που έχουμε τι τροπολογίες με δύο, μετά από δύο εβδομάδες εδώ και ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, γιατί είχα τη δική μου έκθεση και δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή έγκαιρα με τις συζητήσεις. Πάντως ε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να παρουσιάσω. Καταρχήν, Τώρα, ναι. κατά πόσο μπορούμε να πούμε, η τροπολογία να είναι ένα πέμπτο των ε, κρατών μελών ή ένα τρίτο των ε, κρατών μελών είναι τόσο σημαντικό. Ίσως δεν καταλαβαίνω σωστά και τις τροπολογίες. Εγώ βλέπω να υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των τροπολογιών 1 και 10, γιατί μια φορά αναφέρεται ένα πέμπτο των ε, κρατών μελών στην ε, Άρθρο 10 αναφέρεται ένα τέταρτο. Ίσως υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα διατύπωση ή εγώ δεν τα κατάλαβα σωστά τα πράγματα. Ε, εκτός αυτού, όπως και συνάδελφο Μπίλτ, για την... το θέμα της ηλικία συμφωνώ. Και εκτός αυτό πρέπει να εφαρμόσει το δίκαιο των εκάστοτε κράτους μέλους. Στη Γερμανία, στις ε, τοπικές εκλογές η ηλικία των είναι 16. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να επιβάλλουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή κάποιος να μπορεί να συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι σε εθνικό. Αυτό δεν μου φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά όχι δεν είναι και το πιο τεράστιο ε, πρόβλημα. Θα είναι καλό να προσαρμοστούμε. Επίσης, αυτό που είναι σωστό είναι αυτό που αφορά τα και καλυμμένα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα ήταν καλό να έχουμε μια κοινή ιδέα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να, καλύπτει, που να καλύπτεται από όλους. Και τώρα αναφέρομαι σε αρχές ε, και σε αξίες. Ίσως πάμε πάει πολύ μακριά γιατί μπορεί να είναι κάποιες πολιτικές ε, Α παραδείγματο χάρη, ίσως κάποιο κράτο να θέλει να εισαγάγει την θανατική ποινή στην Ευρώπη, Προφανώ όλοι θα είναι αντίθετα, αλλά αν έχουμε κάτι άλλο, όπω την ε, προστασία των μητέρων, ε, αν θέλουμε να ε, εξαλείψουμε κάποιες προθεσμίες προστασίας, αυτό σημαίνει ότι είναι αντίθετο με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχει κάποια πολιτική σημασία. Και εδώ ακριβώς δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο Μπίλτ ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν πρέπει να ξεκινήσουν από εκλεγμένους πολιτικούς. Όχι, και εμείς είμαστε. Κα, κα, κα, είμαστε και εμείς πολίτες και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας να αντιθέση προς τους εθνικούς βουλευτές. Επίσης, εγώ είμαι κατά της μείωσης στα 5.000, γιατί ακριβώς τότε οι Ευρωπαίοι λο, λο, εκπρόσωποι λόμπι, τα συνδικάτα κλπ που μπορούν να κινητοποιήσουν τις 5.000 ανθρώπους ε, θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επίδραση παρά να γενικά σε κάποια ποσοστά κλπ. και θα ήταν καλό όπως προτείνει και η συγκήτρια να υπάρχει ένα ε, σύστημα συλλογής στο διαδίκτυο των υπογραφών έχουμε κάτι παρόμοιο στη Γερμανική Βουλή τέλος δύο παρατηρήσεις ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι σημαίνει η τροπολογία 22 και 26 θέμα του που μένει κανένας και ποια υπηκότητα έχει, είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό όπως υπάρχει εδώ στο κείμενο, αλλά εντάξει να μου το εξηγήσει η συγγήτρια. Και τέλος όπως και στον άλλο Κλάς μπορώ να συμφωνήσω το θέμα της του αριθμού κοινωνικής προστασίας, ε, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε εγώ, μόνο εγώ δεν τον ξέρω κάτω δικό μου τον αριθμό. Θα τον ξέρω έξω. Γιατί υπάρχουν χώρε όπω δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κανένα μία ταυτότητα απάνω του. Δηλαδή, αν με ρωτήσει εμένα σε μια πλατεία και μου ζητήσει υπογραφή μου, θα πρέπει να πάω σπίτι μου και να γυρίσω με, το, με την ε, ταυτότητά μου. Γιατί πολλά στοιχεία ζητώνται εδώ. γιατί μπορεί κανένας μέσω της διεύθυνση να δει κατά πόσο το άτομο αυτό υπάρχει και αν υπάρχει στη διεύθυνση αυτή πραγματικά, αν χρειάζεται. Γιατί η έλλειψη νοστιχίου στοιχείου δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η υπογραφή του. Παραδείγματο, αν κανένα δεν έχει διεύθυνση email, δεν θα πει ότι δεν μπορεί να υπογράψει την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία πολιτών ακούγεται πολύ ωραία. Οι προσδοκίες όντως είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι περιμένουν θαύματα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μαζευτούν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Υπάρχουν πολλά θετικά και έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Για τα 16, την ηλικία των 16. Εγώ πιστεύω ότι τα 18 είναι προτιμότερα. Γιατί από τα 18 ψηφίζουν οι άνθρωποι στις περισσότερες χώρες μέλη. Νομίζω ότι ταιριάζει. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό. Υπάρχει και έκθεση DAF που το λέει. Τώρα, ο πυρήνας του ζητήματος ποιος είναι. Το είπε και ο κύριος Κλάς. Αυτό το θέμα της ε, συγκαλυμμένης αντίθεσης με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βέβαια καθόλου ξεκάθαρο. Το παραδεκτό. Πώς θα κρυθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλά, αν υπάρχει συνθήκη, εντάξει. Αλλά αν υπάρχουν ένα εκατομμύριο υπογραφές, φτάνει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές υπογραφές για να είναι παραδεκτή μια πρόταση. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτό που αναφέρεται σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να ανατρέψουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας τελικά. Δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί εδώ πέρα να περιορίσει αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει από πριν να υπάρχουν τα κριτήρια. άμα θέλουν να ζητήσουν κάτι για την επικουρικότητα οι πολίτες. Ίσως μέσα από τα εθνικά κοινοβούλια να πηγαίνει πιο γρήγορα η διαδικασία, αλλά αν θέλουν να απευθυνθούν σε μας και για την ιστοσελίδα αυτά που είπατε. Να υπάρχει όντως μία ιστοσελίδα. Αλλά προσοχή να μην ε, το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε παραπάνω προπαγάδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να παραμείνει για τη δουλειά που έχει φτιαχτεί και όχι να βάλουμε ένα σωρό πράγματα σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, η κυρία Μιλτσέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πίστευω ότι πρόκειται για ένα μοναδικό μέσο το οποίο πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο για τους πολίτες με και να έχει στόχους απλούς και σαφείς. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής της ομάδας μου και πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει μια συνεκτική θέση για την πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να έχουμε μία ισχυρή θέση έναντι του Συμβουλίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με τις θέσεις ε, των εισηγητριών. Οι δύο εισηγητές ε, της ΑΦΚΟ είπαν ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν φίλτρα στην λήψη απόφασης της Κομισιόν, αλλά να γίνεται σεβαστή μόνο η νομική βάση, ούτως ώστε να μην, οι πρωτοβουλίες πολιτών να μην είναι ε, άτοπες, ε, άστοχες ή ευτράπελες. Να μην έχουμε λοιπόν καταχρηστικές, παράλογες ή αβάσιμες πρωτοβουλίες. Για το θέμα τώρα του εκατομμυρίου των υπογραφών και την κατανομή τους ε, στα κράτη-μέλη και εδώ νομίζω μπορούμε να βρούμε έναν συμβιβασμό. Αλλά πιστεύω ότι αν κρατήσουμε αυτό το φίλτρο που λέτε εσείς 5.000 υπογραφές για το θέμα της, ε, κατά τη φάση της αποδοχής, ε, αυτή η αρχή του ενός τετάρτου κλπ θα πρέπει να εφαρμόζεται και εδώ. Γιατί εγώ μπορώ να ξεκινήσω μία πρωτοβουλία σε ένα χωριό 5.000 κατοίκων και μπορώ πραγματικά έτσι να νοθεύσω το πνεύμα της πρωτοβουλίας των πολιτών, διότι δεν θα είναι πλέον πρωτοβουλία πολιτών. Υποστηρίζω αυτό που είπε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για την διαφάνεια, την οικονομική διαφάνεια και αυτό πρέπει να το εσωματώσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσθέσω τώρα και κάτι άλλο για το θέμα της ταυτότητας. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνουμε τον αριθμό ταυτότητας στο ερωτηματολόγιο υπογραφών. Θα πρέπει να αναφέρεται είτε η υπηκότητα είτε η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Και θα μπορούσε να αποτελέσει και το βασικό κριτήριο. Και δεύτερο, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως δεύτερο κριτήριο την υπηκότητα. Άλλα δύο σημεία. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε στο όριο ηλικίας των ευρωεκλογών, 18 και όχι 16, και θα ήθελα η συλλογή των υπογραφών να περιοριστεί σε ένα χρόνο και όχι σε τέσσερα, διότι τέσσερα πια είναι πολύς χρόνος, πόσο μάλλον για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Και πριν αναφέρθηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξυπνάει τεράστιες προσδοκίες. Αλλά στο κάτω-κάτω αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Να κάνουμε τον κόσμο να μπορεί πιο εύκολα να έχει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μην μειώσουμε τις προσδοκίες, όχι. Να τις διατηρήσουμε. Τουλάχιστον να υπάρχει προστιθέμενη αξία με το μέσο αυτό που είναι η πρωτοβουλία πολιτών. Να είναι κάτι παραπάνω από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα που είναι η διαδικασία αναφορών. Γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιδρούν στις πρωτοβουλίες πολιτών. Να μην λένε ενδεχομένω, αν δεν συμφωνούμε με αυτή την πρωτοβουλία, πάει τελείωσε, τελεία και παύλα. Όχι. Είναι ένα σημαντικό μέσο που θα βοηθήσει οι πολίτες μας να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπόνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Άρα δεν πρέπει να βάζουμε πολύ ψηλά εμπόδια, πολύ μεγάλα εμπόδια, κάθε άλλο. Και για να μπορούν περισσότεροι ακόμα να συμμετέχουν, για μένα το 16 θα έλεγα ότι είναι ήδη μεγάλη ηλικία και όχι μικρή. Αν θέλεις ο κόσμος να νιώθει ότι ανήκει στην Ευρώπη και ότι η Ευρώπη του ανήκει, αυτό πρέπει να γίνεται από νεαρότερη ακόμα ηλικία, όχι τα 16. Οπότε εγώ δεν βλέπω γιατί στα 16 δεν μπορεί ένας νέος να ε, συμμετάσχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία. για την συγκέντρωση υπογραφών. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία. Εξάλλου και η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία του ιδιωτικού βίου ήταν ιδιαίτερα επικριτική στο να μαζεύουμε τόσα συγκεκριμένα στοιχεία. Έπειτα πιστεύω ότι με το που καταγράφεται μία πρωτοβουλία, αμέσω πρέπει να ελέγχεται το παραδεκτό ή όχι. Και όχι πρώτα να συγκεντρώνονται ένα σωρό υπογραφέ και μετά να του λέμε Α, συγγνώμη, δεν είναι παραδεκτή η πρωτοβουλία αυτή. Για την ιστοσελίδα, ναι. Χαίρομαι που συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει μια ιστοσελίδα ανοιχτή πηγή. Και τέλος το 1 τρίτο συμμετοχή δηλαδή πολιτών από το 1 τρίτο των χωρών μελών, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περιοριστικό. Θα πρέπει να λέμε το 1 πέμπτο να φτάνει για να μπορούν περισσότεροι πολίτες και περισσότερες πρωτοβουλίες να προχωρήσουν. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, δημοψηφίσματα σε διάφορες ε, χώρες, αλλά δεν φτάνει. Το θέμα είναι να μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι 48 μήνες ή τέλος πάντων μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να συγκεντρωθούν ε, υπογραφές δεν είναι εφικτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί όχι. Μπορεί πολιτικά να διαφωνεί κανείς, αλλά εγώ δεν βλέπω στην πράξη γιατί να υπάρχει πρόβλημα στο να είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα συγκέντρωσης υπογραφών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βερζέτ Euh, merci, euh, Monsieur le Président. Euh, je suis d'accord avec une grande partie de ce qu'ont dit certains de mes collègues, mais comme il y a... Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τους συναδέλφους, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και μερικές ε, αντιφάσεις. Ο Ντενίς ε, Ζων ήταν υπεύθυνος της ΓΟΕ και ζητά συγγνώμη δεν μπορεί να είναι σήμερα παρόν αλλά συνεργαζόμαστε όμως γιατί εγώ είμαι σάντοου εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτισμού. Η Επιτροπή Πολιτισμού είναι η πρώτη που εργάστηκε γύρω από τον Τοσκέ και επέβαλε προτάσεις ε, σχετικά με την ανάπτυξη της ηθαγένειας και το ρόλο της νεολαίας όλα αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κύριος για το όριο ηλικίας 16 ετών επειδή μία πρωτοβουλία πολιτών δεν έχει νομοθετική απόλυξη εγώ πιστεύω ότι όπως και η Επιτροπή Πολιτισμού το όριο θα έπρεπε να είναι 16 χρονών. Σύμφωνο επίσης και με την τροπολογία για να μειώσουμε το κατόφλι κατά ένα τέταρτο. Τώρα η, πρώτη, η Επιτροπή Πολιτισμού σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτείνει Οργανωτική Επιτροπή εννέα μελών που να ανήκουν στο 1 τέταρτο των χωρών όπως επίσης ε, και η κατάργηση της πρότασης ε, για το κατά πόσο να αποδεκτή όχι πρόταση. Βέβαια θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Πρέπει να αποφύγουμε, να ενισχύουμε την δυσπιστία έναντι των ε, πρωτοβουλειών πολιτών. Θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα σταματήσει να θεωρεί τους πολίτες ως φόβητρα. Θα πρέπει επίσης πιστεύω να δημοσιοποιούνται οι απορρίψεις προτάσεων και η αιτιολόγησή τους. Τώρα για την ιστοσελίδα, ε, εγώ ικανοποιούμε με την απάντηση της Κομισιόν, αυτό τι θέση ανταποκρίνεται και στις θέσεις που εκφράσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά έχω μία ερώτηση σχετικά με αυτήν την συνεχή παραπομπή στα κράτη-μέλη για τους ελέγχους. Γιατί όπως και η Ιντβελ και εγώ και εμένα πραγματικά με καίει το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πραγματική επαγρύπνηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Προστασία δεδομένων και ως προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα εθνικά όργανα και τους οργανωτές. Πρέπει λοιπόν να προστατεύονται οι πολίτες. Έχω απορίες σχετικά με την τροπολογία 4, συμφωνώ δε με την τροπολογία 5. Πιστεύω, όπως και άλλοι είπανε, θα πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση πληροφοριών. Εμείς προτείνουμε ηλικία και τόπο κατοικίας και φτάνει. Και κανένας αριθμός ε, ταυτότητας, διότι Πρωτοβουλία πολιτών δεν σημαίνει ψηφοφορία. Ας σταματήσουμε λοιπόν να είμαστε δύσπιστοι. Είπαμε, πλήρης άρνηση για το δελτίο ταυτότητας. Δεν ισχύει παντού και μπες περιπτώσει δεν χρειάζεται. Επίσης, διαφάνεια απόλυτη για τη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών και των αργωνωτών. Ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού θέλουμε να απομακρύνουμε τους ε, εκλεγμένους αντιπροσώπους από αυτές τις πρωτοβουλίες, όχι γιατί δεν είναι πολίτες οι άνθρωποι, αλλά αυτοί έχουν άλλα κανάλια παρέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι πρωτοβουλίες να είναι καθαρά πρωτοβουλίες πολιτών. Για την προθεσμία 12 μηνών και 48 μηνών έχουμε και τους 6 μήνες Νομίζω ότι είναι όμως αντιφατικό να μειώσουμε αυτή την περίοδο συλλογής των πρώτων υπογραφών και να παρατείνουμε εκείνη του τέλους. Μα εγώ νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι το μάζεμα των 5.000 υπογραφών. Λοιπόν, εγώ είμαι στρατευμένη υπέρ της ηθαγένειας του τόπου κατοικίας και όχι του αίματος. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτήν τη λογική μιλώντας δηλαδή για τους πολίτες κατοικούντες. Ευχαριστώ κυρία Βεργάς. Άλλα σημεία. Κύριος Μπρόγκς. Εγώ είμαι υπέρ ε, της τροπολογίας που στις 300000 300.000-4.000 υπογραφές Είμαι υπέγραφος της τροπολογίας που μειώνει τις τρεις χώρες σε μία και τη μειωσή για το 1 εκατομμύριο από ένα τρίτο το χρόνο στο ένα τέταρτο. Και η διεύρυνση επίση από 12 μήνες σε 48 μήνες για συλλογή των φωτοβουλών και την ιστοσελίδα βέβαια για την συλλογή πληροφοριών. Όλα αυτά μαζί κατά τη γνώμη μου θα επιτρέπουν πραγματικές ε, πρωτοβουλίες των πολιτών να είναι επιτυχείς και όχι εκείνες που οργανώνονται από μεγάλες οργανώσεις. Είμαι κατά της διεύρυνσης των κριτηρίων των ευρωπαϊκών αξιών. Αλλά είμαι κατά γενικά των ε, ε, του κριτηρίου των ευρωπαϊκών αξιών. Θα προσ... τα προστιμούσα μια πιο αυστηρή συζήτηση και περιορισμού για αυτό που μπορούν να εκθούν. Αλλά κύριε Πρόεδρε, αυτό που δίνεται είναι μια ουσιαστική πρόταση, ίσω δεν επιτρέπεται γιατί είναι αντίθετη προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Επιτρέπεται όμως συμπληρωματικά να ζητούμε μία προσθήκη στις ευρωπαϊκές ε, αξίες ή μία διαγραφή κάποιων αξιών ή μία τροποποίηση. Ίσως και αυτό θα ήταν ένα σημείο. Το κριτήριο της ε, αρμοδιότητας είναι το θέμα αρμοδιότητας της Κομισιόν. Όπως το καταλαβαίνω αυτό. Στην ΑΦΚΟ την περασμένη εβδομάδα πολλοί βουλευτές πολύ μάλιστα πολύ γνωστή, είπε ότι ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να προωθήσει αλλαγές στη συνθήκη πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι μπορούν ίσως ευέλικτα να χρησιμοποιήσουν το κριτήριο της αρμοδιότητας προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό αληθεύει ή όχι. Τέλος, η έννοια της δημοκρατίας χρησιμοποιήθηκε και συγκεκριμένα της άμεσης δημοκρατίας. Αλλά όπως ελέγχθη ήδη αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι δημοψηφίσματα, είναι αναφορές που τις αποκαλούμε διαφορετικά. Και μια μάλιστα είναι αναφορές οι οποίες μπορούν να αγνοηθούν εκ μιας αρχής ή να εξαλειφθούν από την Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι άποψε και ε, υπάρχουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές, μην μπορεί να αγνοήσει την αναφορά αυτή η Κομισιόν, αλλά να οδηγηθεί σε ένα δημοψήφισμα. Πρώτος ευχαριστώ. Είχαμε ευρία συζήτηση. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και ευέλικτο. Αν δεν έχουμε άλλες παρατηρήσεις, θα ακούσουμε τους, τις συζήτητες. Η Σεσίλια, η Κίνα, ποιος θα μιλήσει. Παρακαλώ η Σεσίλια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ξέχασα ότι είμαι Σουηδέζα, θα έπρεπε να μιλάω Σουηδικά, διότι έχουμε εξαιρετικού διερμηνείς. Λέει η ομιλήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που πραγματικά <coughs> πάλεψαν σε βάθο. Ε, για αυτήν την ε, έκθεση. Σε αυτές τις σκοτεινές αίθουσες λοιπόν έχει αρχίσει και πνέει νέος άμενεμος, ε, υπάρχει μια σχετική δροσιά. Άκουσα όλους όσους ε, τοποθετήθηκαν. για την καταγραφή των διαφόρων στοιχείων όσο το δυνατόν πιο εγγυημένοι, δηλαδή φυσικά να μην υπάρχουν ούτε φορολογικός, φορολογικός κώδικας, ούτε αριθμοί ταυτότητας, ούτε τέτοια πράγματα. Επίσης πιστεύω ότι είναι εξαιρετική και λογική η πρόταση να μην έχουμε δύο φάσεις στην αποδοχή αλλά μία επίσης αυτό της ηλικίας των 16 ετών. Μα ήταν ο μαγικός αριθμός για να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι. Μα δεν πρόκειται εδώ για την ομοθετική ηλικία. Πρόκειται όμως για μία ηλικία όπου οι νέοι θα μπορούσαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, τις ιδέες τους που θα βελτιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να κατεβάσουμε λοιπόν το κατόφλι για να εμπλακούν οι νέοι. Επίσης το software θα μας το παρέχει η Κομισιόν για την προστασία των δεδομένων. Επίσης θέλουμε να συστήσουμε και μία γραμματεία ε, για τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να ευνοήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών. Ωραιότατες προτάσεις από τους συναδέλφους και χαίρομαι ιδιαίτερα που τις άκουσα και θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν σχετικά. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόντς, θέλετε κι εσείς. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση. Συμφωνώ με διάφορα από τα σχόλια που έγιναν. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε μια γενική ε, πρωτοβουλία των πολιτών που ξεκινάει από τους πολιτές ε, ε, η διαφάνεια είναι επίση σημαντική. Επίση, εμεί δεν τροποποιούμε αυτή τη στιγμή τη συνθήκη τη Λισαβόνα, απλώ δρούμε μέσα στα πλαίσια τη συνθήκη αυτή. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που μπορούμε να αλλάξουν, αλλά έχουμε κάποια ελευθερία να έχουμε την πρόταση αυτή που είναι φιλική προ του πολίτε και συμφωνώ με την κυρία Ντέτσεβα που είπε ότι θα πρέπει να είναι ενιαία η πρωτοβουλία αυτή και να ενωμένο το κοινοβούλιο να την υποστηρίξει. Έχω κάποιες σχέσεις επίσης. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στην ηλικία 16, 18, 17 κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαφορές ε, ε, εθνικές όσον αφορά την ηλικία. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και αυτό είναι το δύσκολο. Κάτι θα πρέπει να έχουμε. Το άλλο σημαντικό που αναφέρθηκε που κλειστά έχεις μάλιστα είναι το θέμα της ε, προστασίας των προσωπικών στοιχείων. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα αναγνωριστούν οι πολίτες και είδαμε ότι σε διάφορα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία για να μπορέσει να οριστεί ένα άτομο. Δηλαδή θα αρχίσουμε με την υπηκότητα και το ελάχιστο των στοιχείων. Αλλά νομίζω η προστασία των στοιχείων είναι ουσιαστικό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ πάλι για την υποστήριξή σας για τις πολύ σημαντικές σας παρατηρήσεις. Και είδατε ότι οι υδροφολογικές ε, μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι. Εκεί λίγη η προθεσμία. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συζήτηση. Και ελπίζω να συμφωνήσουμε και με τις άλλες συναρμόδιες επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους και σας ευχαριστώ για τη συνεχή σας συζήτηση αυτή, την τόσο σημαντική. Και όπως ελέγχθη, η προθεσμία για τις ε, λήγει λίγη αύριο το μεσημέρι στις 12. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 26 Οκτωβρίου, συνεδρία της Επιτροπής μας και στην Ολομέρεια η ψηφοφορία θα γίνει το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λοιπόν να προχωρήσουμε στο σημείο 10. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε πριν να συναντήσουμε σε άλλου από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Το σημείο 10 αφορά την ενίσχυση χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σχετικό σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης από την κυρία Γκόμες όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ορολογικής, πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα που καλύπτει διάφορες πτυχές συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την ανείχνευση και προετοιμασία και αντίδραση. τη χημική καταστροφή στην Ουγγαρία τονίζει τη σημασία του θέματος. Και γι' αυτό θα ακούσουμε σχετικά την εισηγήτριά μας, την κυρία, κυρία Γκόμες. Καταρχήν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως ότι η προθεσμία για την υποβολή προπολογιών είναι μεσημέρι 18 Οκτωβρίου. Η ε, κυρία Γκόμες παρακαλώ. Mr. President, um, I wish to, first uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν ήδη γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή Βιομηχανίας, ΝΑΦΕΤ και από την Επιτροπή Επιτροπή Ένβη που συνέβαλε πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρώτη φορά που εξετάστηκε το θέμα αυτό βιολογικών, ρεδιολογικών και πυρηνικών μέσων ήταν μετά τις επιθέσεις της 9 της 11 ε, Σεπτεμβρίου. Αυτό το πρόγραμμα δράση που αφορά την έκθεση υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο 2009 πριν τεθεί σε ισχύ δηλαδή η συνθήκη και βάσει σε μια ανακοίνωση κομισιών ε, από τον Ιούνιο του 2009. Η εξολόγηση δική μου του προγράμματος δράσεως με έκανε να πιστεύω ότι το σχέδιο αυτό έχει μειώσει σημαντικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Η συστάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι να επανενδυναμώσουμε τις διάφορες πτυχές αυτές που έχουν αποδυναμωθεί από το Συμβούλιο. δεν εξετάζουμε μονάχα για τα δυστυχήματα χ, β, αλλά και πραγματικά δυστυχήματα που οφείλουν σε ανθρώπινο σφάλμα, όπως αυτό που αυτή τη στιγμή έλαβε χώρα στην Ουγγαρία. χημική καταστροφή. Και μέσα στο νέο πλαίσιο μέσα στη νέα δεσμένη αρμοδιότητα που απαραίει από τις συνθήκες Λισαβόνας, θα πρέπει να έχουμε καλύτερο συνδυασμό μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν και μεταξύ διαφορών θεσμικών οργάνων, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε το θέμα της πρόληψης, το θέμα της ανείχνευσης και το θέμα της ανίδρασης. Επίσης είναι σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μη, ένας δημοκρατικός έλεγχος. Το σημαντικό είναι αυτή, η, αυτός ο συγχαρισμός των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του κινδύνου χιβιταροποίηση. Χρειάζεται αναλυτική παρουσίαση, κοινό προγραμματισμό, ανάπτυξη μεθόδων αντίδρασης, αποτελεσματική χρήση των υπερχόντων πόρων κλπ. Παραδείγματο χάρη, οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Περιβάλλοντο είπαν ότι η αντίδραση των κρατών μελών στην ε, πανδημία του H1N δεν ήταν συντονισμένοι. Δηλαδή τα κράτη-μέλη συνέντευξαν μη συντονισμένα. Ο καθένα έκανε ό,τι νόμιζε ότι ήταν καλύτερα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι όταν εξετάζουμε την ανάγκη εποπτείας από το κοινοβούλιο αυτό εδώ και τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με τη συνθήκη της Δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν συζητάμε για τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Αλλά τα δυστυχήματα αυτά δεν σέβονται τα σύνορα. Είναι μεθοριακά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ανάλογη προσέγγιση. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η αντίδραση και η προετοιμασία για αυτού του τύπου τα δυστυχήματα προσφέρει τη δυνατότητα στα κρατημένη και στην Κομισιό να πραγματοποιήσουν συνθήκη αλληλεγγύης που ήδη υπάρχει στην σύμβαση της συνθήκης της Αλλά δυστυχώς η, η συμφωνία που υπάρχει, το σχέδιο δράσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν προβλέπει τη χρήση της ρήτρας αυτής αλληλεγγύης. Για να είμαι σύντομη, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω απλώ να τονίσω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατεπηγόντως ένα μηχανισμό ευρωπαϊκό αντίδρασης που θα ειδικεύεται σε αυτού του τύπου τα δυστυχήματα. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια δυνατότητα συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών οργανώσεων και υπηρεσιών. Γιατί και οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν πάρα πολλές γνώσεις και δεν μπορούμε να τις εγνοήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που δίνει δυνατότητα στην Ουγγαρία να αντιμετωπίσει αυτό το χημικό δυστύχημα και θα ήθελα αυτή η νέα υπηρεσία πολιτικής προστασίας που υπάρχει από την εποχή της έκθεσης Παρνιέ θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με τις στρατιωτικές υπηρεσίες που έχουν πάρα πολύ εμπειρία στην πρόληψη, στην ανείχνευση των δυστυχημάτων αυτών. και επίσης η αντίδραση με τις υπηρεσίες ε, αντικατασκοπίας, τις υπηρεσίες ε, δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική και εδώ επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και η δική μας κοινοβουλευτική εποπτεία. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι ο συντονιστής αντιτροποκριτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι υπόλογος κλπ. Εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, ε, κοιτάζω ποιες είναι οι επιπτώσεις στα μέσα εξωτερικών δράσεων και η σχέση με τη βιομηχανία. Γιατί αυτά τα υλικά είναι υλικά που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ουγγαρία. Γι' αυτό αναφέρομαι στην ανάγκη τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν να αντιταχθούν στις προτάσεις της βιομηχανίας να μην υπάρχει τόση πολλή νομοθεσία διακανονισμού. γιατί το λέμε ότι θα πρέπει να έχει διακονιστικές αρμοδιότητες η Κομισιόν για να μπορεί να παρακολουθεί και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κανονισμών. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η εφαρμογή των ε, συνθήκων και η αποφυγή της καταπάτησης αυτών. και πρέπει να δούμε επίσης ε, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, ε, τα χρονικά διαστήματα, προθεσμίες να υπάρχουν ε, επιτόπου προετοιμασίες εκάστοτε σε όλη την επικράτεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι παρόμοιο προτείνει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των προβλημάτων. Όπως είπε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι πολιτικές υπηρεσίες που είναι οι πρώτοι εταίροι στην περίπτωση όταν υπάρχουν αυτά τα και βιολογικές όπως ο άνθρακας ε, οι χημικές δεν αρκεί όπως είναι προετοιμασμένες. Θα πρέπει να είναι έτοιμες σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι ειδικευμένε. Να δίνουν το προσωπικό, ιατρικό προσωπικό και έτσι οι υπηρεσίες πολιτικές και στρατιωτικές να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις απειλές. Και εν τελευταία αναλύση είναι να φροντίσουμε το Συμβούλιο να προωθήσει το πρόγραμμα δράσης, να το καθαστήσει πιο ισχυρό και να φροντίσει και το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορούν να ασκήσουν όλες τους αρμοδιότητες στο τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκόμες. Η Προεδρία, η Κομισιόν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Όχι. Δεν ενδιαφέρονται. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Ε, οι συνάδελφοι, η κυρία Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την εξαιρετική της συνεργασία. Στόχος μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές είναι ο στόχος μας για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές είναι κάτι το οποίο εγώ συμμερίζομαι. Πρέπει πραγματικά αυτές τις απειλές να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι το Συμβούλιο τα ενέκρινε όλα αυτά εν απουσία του Κοινοβουλίου. Και εμείς εδώ γνωμοδοτούμε ένα χρόνο μετά από την έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο. Τέλος πάντων, καλυρούμε να δώσουμε και εμείς καμία πρόταση ευφυή προς το Συμβούλιο για να διορθώσει κάπως τα πράγματα. Θέλουμε έναν καθαρότερο ρόλο μεταξύ των όσων εφαρμόζουν το σχεδίο. Ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός και από στρατιωτικής πλευράς και από πολιτικής πλευράς. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός. Πρέπει να εφαρμόσουμε όσο είναι δυνατόν τις ήδη υπάρχουσες υποδομές. και η δημιουργία νέων υποδομών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο όταν αυτές οι υποδομές που έχουμε είναι ανεπαρκείς. Έχω μία τροπολογία λοιπόν. Όσον αφορά στα αντίδοτα, θα πρέπει να έχουμε αποθέματα. Σε περίπτωση βιολογικών επιθέσεων, είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να συνεργάζονται ούτως ώστε να έχουμε αποθήκες τέτοιες οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν σε μία μαζική επίθεση. Αυτά τα αποθέματα που έχουμε σήμερα δεν είναι επαρκή. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τον αριθμό τους. Χρειάζεται λοιπόν σοβαρότητα στην προσέγγιση μας, εκφράζουμε όπως είπε και η συγγήτρια τη λύπη μας ε, για το γεγονός ε, της ε, τελευταίας αυτής καταστροφής στην Ουγγαρία με όλη αυτή την τραγωδία τέλο πάντων στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες πρέπει λοιπόν να εργαστούμε το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την εισηγήτρια και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά στη χημική βιομηχανία όταν ε, ε, σχολίασε ότι η χημική βιομηχανία κάποιες φορές αναφέρει ότι η πολλή νομοθεσία δυσχεραίνει το έργο της. Νομίζω και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ στη συζήτηση ότι ειδικά στο θέμα της, προ... της πρόληψης δεν πρέπει να κάνουμε καμία έκπτωση αν υπάρχει κάποια νομοθεσία την οποία πρέπει να κάνουμε όσο πιο ισχυρή γίνεται και να δώσουμε έμφαση είναι εκείνη που αναφέρεται στην απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου. Ε, συζητάμε την αντιμετώπιση, συζητάμε τη διαχείριση, συζητάμε το μηχανισμό που πρέπει να έχουμε. Αν μη τι άλλο όμως, αν θέλουμε μεσοπρόθεσμα να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και οι λύσεις που θα προωθήσουμε να είναι τελικά πιο αποτελεσματικές και από την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο του 2009, ε, νομίζω ότι η πρόληψη είναι ε, μια αφετηρία πολύ σημαντική. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και σε αυτό το θέμα, εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας, του Ευρωπαϊκού, του EPP, να παρακαλέσω να παραταθεί η προθεσμία για τις τροπολογίες, διότι επαναλαμβάνω και πάλι αυτή η εβδομάδα σχεδόν ε, όλοι οι συνάδελφοι θα λείπουμε στην, Πορτογαλία και μέχρι την Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά που είναι η προθεσμία, δεν θα μπορέσουμε έγκαιρα να εργαστούμε όσο αποτελεσματικά θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Δίας Δεμέρα. Πρόσι υπογράφω το όσα είπε ο συνάδελφος Παπα-Νικολάου. Ούτως ώστε να παρατείνουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και θέλω να κάνω μία δήλωση. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ ευρύ, μεγάλο. Μιλάμε εδώ για ένα σχέδιο δράσης. Για να αντιμετωπίσουμε κινδύνους, απειλές, αντιδράσεις, επιπτώσεις, αποθεομηνίες... ή καταστροφές που προκαλούν οι διεστραμμένοι άνθρωποι. Μιλάμε λοιπόν για το χημικό, το βιολογικό και το ραδιενεργό. Πρόκειται για ένα τεράστιο φάσμα. Η πρώτη δήλωση λοιπόν που κάνω είναι ότι είμαι σκεπτικιστής για την αποτελεσματικότητα ενός ε, τόσο ευραίος ε, ε, ε, πεδίου δράσης. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πρώτα την πρόληψη και μετά την αντίδραση. Και αυτού του είδους δε οι καταστροφές έχουν ε, διεθνικό χαρακτήρα. Δείτε τι έγινε με την Ουγγαρία. Αυτή η, αυτή καταστροφή θα πλήξει τέσσερις χώρες μέσα από το, από το Δούναβι. Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση, να την εμπλουτίσουμε με τροπολογίες και να προβληματιστούμε ιδιαίτερα για το τι εστί πρόληψη και το τι εστί αντίδραση. Μπορούμε να φιλοσοφήσουμε για την πρόληψη και σίγουρα μπορεί να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω και το βέω δηλαδή, το, το, από την εμπειρία μου το βλέπω δυστυχώς, το βλέπω δύσκολο και πολύ πλοκό να έχουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης σε αυτούς τους τομείς, γιατί η αντίδραση είναι τρία πράγματα. Αντιδρώ τι σημαίνει, εκενώνω, βοηθώ, καταστέλω. Βασικά αυτή είναι η αντίδραση. Και μετά πρέπει να λάβουμε δύο διαφοροποιημένα πράγματα υπόψη μας. Προστασία των προσώπων και προστασία των υποδομών και των κριτικών υποδομών. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που θα θέλαμε από το ΕΛΚ να τα συζητήσουμε με περισσότερο χρόνο. Τώρα, χειροκροτώ με συμπάθεια τα σχόλια της εισηγήτριας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη σημασία αυτών των τριών-τεσσάρων τομέων που εντάσσονται στην απάντηση στρατιωτικό, αστυνομικό, υγειονομικό και την πολιτική προστασία. Γι' αυτό λοιπόν κυρία μου σας εμψυχώνω να συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση, σας υποστηρίζω και θα φροντίσω να κάνω τροπολογίες έγκαιρα, να υποβάλω έγκαιρα τροπολογίες για να εμπλουτίσουμε αυτή την έκθεση που τόσο χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Διέζη Δεμέρα. Κύριε Μούλτερ θέλετε το λόγο. Ναι, Πάντα, Πρόεδρε. Βλέπετε με θαυμασμό ακούω, γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα πολύ καλά. Βλέπω ότι εδώ μιλάμε για το ρόλο της Επιτροπής και αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί ο κεντρικός ρόλος δεν μπορεί να είναι παρά ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο. Με εκπλήσει επίσης κάπως, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ακρόαση και είχαμε από την Eurojust και την Europol παρεμβάσει, και αν τις κατάλαβα καλά, θεωρούν ότι και εκείνε έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της τρομοκρατίας. Και τα δύο αυτά όργανα λογοδοτούν προς την Επιτροπή. Οπότε η Επιτροπή πρέπει να δίνει συνέχεια. Το βασικό στην έκθεση αυτή λοιπόν είναι ποιο ακριβώ είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε. Κύριε Άλβαρο, αλλά βλέπετε περνάει η ώρα, οπότε βοηθήστε μας να επιταχύνουμε λιγάκι παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί πέρα από την καλή δουλειά που κάνει η Άννα, έχω μια ερώτηση πώς λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα που έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε ένα σύστημα όπως ε, στο Ρίτσο που η κάθε χώρα έπρεπε να δίνει ό,τι στοιχεία έχει. Δεν είναι μια επιπρόσθετη αξία αυτό. Για να ξέρουμε τι επικίνδυνα χημικά κυκλοφορούν, που βρίσκονται και για την πρόληψη και για να μπορούμε να αποφύγουμε πράγματα όπως αυτά που είχαμε στην Ουγγαρία. Δηλαδή και από την ομοθεσία που είχαμε κατά το παρελθόν να κρατάμε τα στοιχεία και το κάθε κράτος να μπορεί να δίνει. Ο κύριος ε, Δεμέρα. Τηλεγραφικά. Να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Μούλτερ. Άννα, θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον να λάβεις υπόψη σου τα δεν είναι μόνο συντονιστής ε, της ε, καταπολέμησης και της τρομοκρατίας ο οποίος θα πρέπει να επισημαίνει τον κίνδυνο, την απειλή, την πρόληψη. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί οργανισμοί που το καταλαβαίνουν αυτά. Europol, Eurojust, ε, ο συντονιστής Καλύτερος λοιπόν από όλους, όπως είπε και ο κύριος Μίλτερ, θα ήταν η Κομισιόν. Η κυρία Αναγκόμε για να ολοκληρώνει. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για τόσα είπαν. Συμφωνώ και εγώ ότι νέος οργανισμός χρειάζεται μόνο όταν είναι αναγκαιότητα. Πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τους ήδη υπάρχοντες ευρωπαϊκούς ε, μηχανισμούς προστασίας. Άπαξ. Και υπάρχουν ε, νέες δυνατότητες. Εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο στη χημική βιομηχανία. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια που ασχολούνται με βιολογικούς παράγοντες, παθολογικούς παράγοντες ναι, πρέπει να γίνει μνήα της οδηγίας για το REACH. Πάντως, ένα σχέδιο δράσης είναι για να δούμε πώς τίθεται σε εφαρμογή, πώς λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες αυτές για το συγκεκριμένο σκοπό. Και τι είδαμε με την Ουγγαρία, μόλις διάβασε ένα σχόλιο. Ότι ασχολούνται με τα πόβλητα των εξορυκτικών βιομηχανιών, αλλά αγνοούν άλλες περιπτώσεις όπως αυτή που είχαμε. Αλλιώς θα είχε αποφευθεί αυτό το ατύχημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε οι οδηγίες που ήδη υπάρχουν, το REACH, τίθεται σε εφαρμογή, το σέβονται οι χώρες, οι χημικές βιομηχανίες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Δίεθ Ντεμέρα. Πράγματι, είναι ένα τεράστιο σχέδιο. Καταλαβαίνω τον σκεπτικισμό του. Αλλά είναι καλύτερο αυτό που κάνουμε, που πάμε βήμα-βήμα, από το να μην κάνουμε τίποτα. Και τελειώς κάποιες χώρες κάτι θα μπορέσουν να κάνουν, πολλές, άλλες μηδέν, δεν θα έχουν τίποτα εφόσον έχουμε να κάνουμε με ατυχήματα ή με επιθέσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα, πρέπει να αναπτύξουμε δυνατότητες αντιμετώπισης τους και να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα το οποίο να διαρθρώνει τις δυνατότητες που έχουν οι χώρες μέλη μεταξύ τους. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κεντρική σημασία, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει δυνατότητες και να προλαμβάνει και να συντονίζει. Πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν ρυθμιστικό, συντονιστικό ρόλο, να μπορεί να συντονίζει όλα αυτά τα όργανα, όπως είπατε κι εσείς. Ακόμα και μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Χρειάζεται μια σωστή διάρθρωση των διαφόρων υπηρεσιών μεταξύ τους. Όσον αφορά για τις προτάσεις για τροπολογίες, ευχαρίστω δεν έχω καμία αντίρρηση, έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Γκόμες. Για να αναβληθεί προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, όπως ζητήθηκε από το ΕΛΚ, καμία ομάδα δεν είχε αντίρρηση. Οπότε προτείνουμε να αναβάλουμε για 15 μέρες την προθεσμία που είχε καθοριστεί αρχικά για τη 18η Οκτωβρίου. Άρα μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι, έχουμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση αυτή. Σύμφωνοι? Αλλά διατηρούμε την ίδια ημερομηνία για να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Όχι, όχι, ε. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία για ψηφοφορία. Κύριε Γκόμες, όπως είπα και οι συνάδελφοι, είναι ένας χρόνος αφού υιοθετήθηκε το σχέδιο πλαίσιο. Μην καθυστερούμε παραπάνω να εγκριθεί στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο παρακαλώ και να πάει στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Θα είναι ένας χρόνος αφού έχει περάσει. Μην περιμένουμε παραπάνω. Για να δούμε. Αν συμφωνήσουμε με το αίτημα που είναι να παρατείνουμε την προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, είναι αναπόφευκτο να πάμε τον Νοέμβριο για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Είναι λογικό. 15 μέρες καθυστέρηση είναι νομίζω λογικό. Κάποια στιγμή με τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου ίσως, να προβλέψουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, οπότε θα μπορούσε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου η έκθεση αυτή. Άρα, έτσι καλώς συνεδριάζουμε τέλη Νοεμβρίου. Η ΛΥΜΠΕ, 26 νομίζω Νοεμβρίου, κάτι τέτοιο. Θα φροντίσουμε τότε να μπει για ψηφοφορία. Εδώ το θέμα αυτό, οπότε να περάσει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Για να επιταχύνουμε λίγο το βήμα μας, γιατί έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ένα από αυτά, μάλιστα, το τελευταίο, είναι και αρκετά ουσιώδες. Οπότε βοηθήστε μας να προχωρήσουμε κάπως πιο γρήγορα για να προλάβουμε και να μην αφήσουμε τους Πολωνούς να μας περιμένουν. Εξήμιση πρέπει να έχουμε τελειώσει. Πάμε λοιπόν τώρα στο σημείο αριθμός 11, που είναι η τροποποίηση του κανονισμού περί καταλόγου τρίτων χωρών, η υπήκοη των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Η συγητής είναι ο συνάδελφος Δίαθ Ντεμέρα. Γνωρίζετε ότι έχουμε ασχοληθεί και άλλη φορά με το θέμα αυτό και έχουμε ακούσει από τον κύριο Δίαθ Ντεμέρα. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Και σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι για αύριο 12 το μεσημέρι. 12 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην ΛΥΜΠΕ στις 26 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια στην Σύνοδο του Νοεμβρίου. Παρακαλώ κύριε Διευθυντεμέρα, Μέρα, έχετε το λόγο. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που το συζητάμε αυτό το θέμα. Ο κανονισμός 539 ε, του 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών που ον οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θεώρησης. Τώρα η πρόσφατη απόφαση για τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Αλβανία όπως επίσης και τις πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίες του Μαυροβουνίου και της Σερβίας του 2009 αποτελούν και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν έχουμε αυτή την πρόταση του κανονισμού και έχουμε σήμερα έναν τριπλό στόχο. Θα σταθώ όμως στους δύο. Για το να βάλουμε την Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο και τα νησιά Μαριάνες. Ε, οι Βόρειες Μαριάνες, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι είναι Αμερικανοί πολίτες οι κατοικοί τους. Ε, ε, έτσι λοιπόν η εξαίρεση αυτή δεν είναι μέτρο απλώς, είναι ε, πολιτική συνάφεια. Τώρα για την Ταϊβάν. Εδώ χρειάζεται μελέτη από την μεριά μου. Η Ταϊβάν έχει προχωρήσει πολύ δημοκρατικά κλπ. Από το 96 έχει δημοκρατία. Οι πρώτες εκλογές, οι πρώτες προεδρικές εκλογές ε, θα γίνουν τη χρονιά που μόλις ανέφερα. Ο πρόεδρος εκλέγεται για τέσσερα χρόνια και ο διορίζει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μετά διορίζει την κυβέρνηση και τα διάφορα υπουργεία. και υπάρχει και η Βουλή με 113 βουλευτές ε, που εκλέγονται με ένα εκλογικό σύστημα ε, ε, χωριστό. Πολύ σύντομα σας τα λέω τώρα αυτά. Η Ταϊβάν είναι από, τα πλουσιο, από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου 35.000 δολάρια κατά κεφαλή Η οικονομική ανάπτυξη ήταν 13,27 κατά το πρώτο εξάμεινο του 2010 και το εμπορικό ισοζύγιο είχε ένα πλεόνασμα 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, 0,15% είναι το ποσοστό μετανάστευσης. Λοιπόν, είναι χαμηλότατη η πιθανότητα να έρθουν μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ταϊβάν. Και μεταξύ 2006-2008 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μόνο 45 παράνομους Ταϊβανέζους. Βλέπετε λοιπόν αμεληταίες ποσότητες. Τώρα για την ασφάλεια κλπ. Πρέπει να σας πω ότι τα ηλεκτρονικά, ε, τα ιβανικά διαβατήρια ενσωματώνουν όλες τις προδιαγραφές της ΙΑΤΑ, όπως επίσης και άλλες σύγχρονες διατάξεις κατά της πλαστογραφίας. Εγώ προσωπικά το διαπίστωσα αυτό. Ή τα Ιβανέζικη διασπορά, κάπου 60.000 άτομα, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή την πρόταση. Πρόκειται για άτομα που έχουν ένα ταϊβανικό διαβατήριο και πρέπει λοιπόν να τους ε, επιτρέπεται η πρόσβαση. Και το ίδιο κριτήριο δηλαδή θα πρέπει να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω και στην έκθεσή μου. Σήμερα η Ταϊβάν δεν απαιτεί βίζα σε 25 χώρες από τις 23 της Ένωσης, εκτός δηλαδή Κύπρου, Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Οι ταϊβανικές αρχές όμως δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην απόλυτη εξαίρεση θεώρησης για την Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία πριν από τα τέλη του 2010. Είπανε λοιπόν οι αρχές της Ταϊβάν που είναι εδώ και παρούς στην αίθουσα και τις χαιρετίζω μας είπαν 11 Νοεμβρίου. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά πείτε το και γραπτά στην Κομισιόν και ορίστε με την Κομισιόν ότι δεσμεύεστε σχετικά γραπτός. Τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία εξαίρεσαν για όλους αυτούς τους λόγους που σας προανέφερα τον Ιούλιο του 2009 τους Ταϊβανούς από την υποχρέωση της θεώρησης και άλλες χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη και Νέα Ζηλανδία έκαναν το αυτό. Και τελειώνω τώρα κύριε Πρόεδρε. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα παράνομης μετανάστευσης από την Ταϊβάν, ούτε θέματα δημόσιας τάξης. Η απολευθέρωση των θεωρήσεων με την Ταϊβάν θα εμπλουτίσει τις σχέσεις της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ευνοήσει μια αμεσότερη συνεργασία για το περιβάλλον, την παιδεία, την κουλτούρα κλπ. Και θα επιτρέψει και την αμοιβαία τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξαιρέσουμε την Ταϊβάν από την θεώρηση. Διότι αυτή η εξαίρεση ισχύει για, τους, για το Μακάο, Χονγκ Κόνγκ, Ιαπωνία, Νότιο Κορία, Σιγκαπούρια. Λοιπόν, ή τα Ιβανέζοι της Διασποράς που έχουν διπλή υπηκότητα και είναι κάπου 60.000 άνθρωποι, αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού διαβατηρίου ούτε του να μπει ο αριθμός ταυτότητας μέσα σε αυτό το διαβατήριο. Αλλά έχουν δύο υπηκότητες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συνάψουμε τις ε, σχέσεις μας και να θεωρήσουμε τις βίζες με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ κύριε Δίδε Μέρα. Τώρα, μήπως η Κομισιόν θέλει να απαντήσει. Εάν δεν αισθάνεται απόλυτα υποχρεωμένος να απαντήσετε και να αντιδράσετε, θα έλεγα να στραφούν προς τους Βουλευτέ που έχουν ζητήσει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κομισιόν που δεν παίρνει το λόγο γιατί έχουμε περιορισμούς χρονικούς. Γιακολίνο, Sentiamo dal nostro collega della... θα είμαι κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την εξαντλητική παρουσίαση και ακριβέστατη ε, παρουσίαση του κυρίου Δεμέρα ο οποίος μας λέει ότι αυτή η επιλογή είναι πλέον, αποτελεί πλέον για μας καθήκον. 60 χρόνια, τα τελευταία 60 χρόνια η Ταϊβάν αναπτύχθηκε όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά και εμπορικά. Αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα, σίγουρα υπάρχει μια πραγματικότητα ε, στην οποία, για την οποία η Ευρώπη τρέφει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια περιοχή όπου η Ευρώπη ξεχωρίζει γιατί δεν ζητάει από τις όμορες χώρες βίζα. Ξεχνάμε όμως κάτι, ότι την Ταϊβάν δεν την έχουν αναγνωρίσει όλες οι χώρες. Το ότι τίνουμε εμείς χείραν στην ε, Ταϊβάν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εγώ πήγα πρόσφατα στην Ταϊβάν, υπάρχει μεγάλη δημοκρατική συμμετοχή, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλίου. Εγώ έχω τη γνώμη ότι αυτό το ντοσία πρέπει να περάσει όσο το δυνατόν σύντομότερα με την έγκριση ενός μέτρου που θα επιτρέπει την δυνατότητα σε πολλούς Ταϊβανέζους να αισθάνονται λιγότερο μονάχοι τους και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ όλους να είναι σύντομοι. Αρχίζω με την κυρία Τάνια Χαντζόν. Ε, εγώ ευχαριστώ τον ε, κύριο Διές Δεμέρα για την εξαντλητική του έκθεση. Εγώ ως και όλες οι συγγήτρες συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της χορήγησης θεωρήσεων είναι απόλυτα λογικό για την Ταϊβάν. Εμείς ε, Είδαμε την εμπειρία, ποια εμπειρία έχουμε με την κατάργηση των θεωρήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε και ένα μέτρο, ένα παρεμφερές μέτρο για την Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Αλβανία. Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών. Απ' την άλλη όμως ενισχύει και την προσαρμογή των τρίτων χωρών στα ζητούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την ε, συνοριακή ασφάλεια. Φυσικά η Ταϊβάν δεν είναι μια επικίνδυνη χώρα, δεν αντιπροσωπεύει κανέναν κίνδυνο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ταϊβάν και θα διευκολυνθούν οι σχέσεις, οι εμπορικές μας σχέσεις με την κατάργηση της βίζας. Υπάρχει και αυτή η αρχή αμοιβαιότητας, όπως λέγαμε 24 χώρες δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης για την Ταϊβάν, ελπίζουμε άλλες τρεις χώρες να μπουν στη λίστα, πρόκειται λοιπόν για μια ανταλλαγή διπλής κατεύθυνσης για την μετανάστευση. Σίγουρα δεν έχουμε το ρίσκο της παράνομης μετανάστευσης διότι δεν έχουμε ανησυχητικά στοιχεία σχετικά. Δηλαδή με τα παράνομη λαθρομετανάστες από την Ταϊβάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν τον συνάδελφο, ο κύριος Άλβαρο. Φυσικά πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Γιατί δεν έχω τίποτα να προσθέσω στην έξω κυρία που τον έχει λεχθεί η Ταϊβάν που γνωρίζω εγώ προσωπικά είναι ακριβώ όπω την περιγράφετε στην έκθεσή σα. Αλλά μια που ασχολείται η έκθεσή σα και με τρίτε χώρε οι οποίε των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίου, όχι μόνο η Ταϊβάν, θα ήθελα να το πω, εδώ δεν ξέρω, κάπου πρέπει να το μας απασχολήσει ω ε, ε, επιτροπή. Δηλαδή τα προγράμματα ε, μη υποχρεωτική βίζα δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για να φοβήσουμε άλλε χώρε. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό να χρησιμοποιείται σαν ένα πολιτικό μέσο να λέμε ότι αν εσείς δεν μας υποστηρίξετε για κάποια θέματα τότε εμείς η Αυστρία Φερρυπίν, θα άρει την ε, απελευθέρωση από θεωρήση διαβατηρίου για τους υπουργούς. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχουμε καμία γενική έκθεση εδώ. Ίσως κύριε στη Μέρα, μήπως ξέρετε που μπορούμε να εκφράσουμε κάποια τέτοια κριτική έναντι εκείνων των εταίρων μας που χρησιμοποιούν την απελευθέρωση από τη Βίζα ε, σαν ένα μέσο για να πετύχουν κάποιου πολιτικού στόχου. Δεν ξέρω, ίσω θέλετε να το βάλετε εδώ όσον αφορά την εκθέση για την Ταϊβάν. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο και θα σα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Τελικά σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Δία Δεμέρα για την εξαιρετική δουλειά του. Ένα σχόλιο μόνο σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν ε, έχω την ενημέρωση ε, από όσα έγγραφα έχω ε, ενώπιόν μου ότι η Ταϊβάν μέχρι το τέλος του 2010 αναμένουμε να μας κοινοποιήσει επίσημα ότι αντιστοίχως έχει άρει την υποχρέωση θεώρησης για τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία, το συνημειώνουμε αυτό. Κύριε Διαθεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ στους τέσσερις συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Ευχαριστώ και την Τάνια Φαγιόν για την ε, υποστήριξή της και τη δέσμευσή της όλη αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ και τον Σαλβατόρε για τη βοήθειά του. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον Σαλβατόρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Παπα-Νικολάου Ευχαριστώ και σένα, Αλεξάνδερ, για την υποστήριξή σου στην έκθεση. Μερικά σχόλια, Αλεξάνδερ, πρόκειται για κοινοβουλευτική ευρότητα. Έχουμε το τομπάγκο σαν τα Λουθία, Γρένα, Δίνες κλπ. κλπ. Αυτές τις χώρες τις έχουν, με προτείνει, έχουν μία ή δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Τώρα για το τελευταίο θέμα πρέπει να κάνουμε μία σημαντικότατη διευκρίνηση για την εξαίρεση θεωρήσεων. Δεν έχουμε εδώ καμιά διμερή συμφωνία. Έχουμε μία μονομερή απόφαση των 27. Γιατί. Διότι η Ταϊβάν έχει εξαιρέσει από θεώρηση 24 χώρες και από ό,τι μας λένε, που θέλουμε να μας το πούνε και γραπτός δηλαδή, πριν από τις 11 Νοεμβρίου θα υπάρξει εξαίρεση θεώρησης και για, για όλους τους 27. Δεν έχουμε εδώ καμία σύμβαση. Πρόκειται για μονομερή απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο κύριο Διέσδε Μέρα, μιλώντας προς τα πίσω και όχι στο μικρόφωνο του. Ευχαριστώ κύριε Διέσδε Δεμέρα. Σημειώσαμε προσεκτικά την πρότασή σας. Η προσωπία του ΔΕΒΑ θα ε, πρέπει να μας κοινοποιήσει την βούλησή της να εντάξει τα τελευταία τρία κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή δεν εξαιρούνται από την ανάγκη θεώρησης. Και βέβαια δεν έχουμε εδώ μία συμφωνία, μία αμοιβαία αντιμετώπιση, είναι μία έκφραση βούλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί η Ταϊβάν στον κατάλογο των χωρών που, τον οποίο οι υποκοί εξαιρούνται τις ανάγκες θεώρησης όταν έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το κατανοούμε αυτό, εντάξει. Και το τελευταίο θέμα που έχουμε είναι, ε, εδώ να μην ξεχάσω να σας πω ότι η προθεσμία είναι αύριο το μεσημέρι στις 12 για τις τροπολογίες και περνάμε, λέω, στο τελευταίο θέμα αυτής της τόσο βεβαρημένης ημερησίας διάταξης Και πρόκειται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Mm. Να ακούσουμε αμέσω τον εισηγητή, τον κύριο Σάμα Μπουσούτη, για την τροπή του κανονισμού που σε 15 του Ευρωπαϊκού για διαχείριση υπηρεσιακή συνεργασία στα κρατικά σύνορα των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Frontex δηλαδή. Ξέρετε ότι η Κομισιόν δημοσίευσε μια πρόταση το Μάρτιο του 2010 για το θέμα αυτό και μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επισκέφθηκε πριν από δύο εβδομάδε στην Frontex στη Βαρσοβία στη Πολωνία δηλαδή και συζήτησε τα θέματα αυτά και με εθνικά κοινοβούλια από την ευκαιρία τη διακοινοβουλική συνάντηση στι 4 Οκτωβρίου. Ο κ. Μπουζοτήλ τώρα θα μα κάνει παρουσίαση έκθεσή του και μετά νομίζω θα μπορέσουμε να ακούσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ κύριε Μπουζοτήλ, να είστε και εσείς Σε Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Πρόκειται για ένα νομοθετικό ζήτημα και έχουμε στη διάθεσή μας 10 λεπτά, ούτε καν 10 λεπτά για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πρόθεσή μου αρχικά ήταν να σας παρουσιάσω στην επόμενη συνεδρίαση το πρώτο γραπτό μου κείμενο τον Οκτώβριο αλλά χωρίς ανταλλαγή απόψεων σήμερα πώς θα το κάνω αυτό. Οπότε θέλω να ρωτήσω τους οι συζητητές Τι προτιμούν. Θέλουν να δεχτούν αυτή τη σημερινή συνάντηση σαν ανταλλαγή απόψεων ή να έχουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Γιατί... Πώς να προλάβουμε. Ρωτάω λοιπόν τους συναδέλφους μου, τους σκιώδες εισηγητές, να με βοηθήσουν να αποφασίσω. Θέλω να έχω την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μια συνάντηση με τους σκιώδεις, αν πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αλλά από την άλλη δεν θέλω να τους κάνω να νομίζουν ότι προσπαθώ να πιέσω και να προχωρήσουμε γρήγορα. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η συνάντησή μας θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, οπότε θα σταματήσω και ζητάω από τους σκιώδεις να πούν τη γνώμη τους παρακαλώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πουσότελ, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε, πράγματι. Συμβαίνει συχνά να έχουμε πάρα πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις μας. Έγινε λοιπόν μία πρόταση. Μήπως μπορούμε να αναβάλουμε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ίσως μπορούμε να ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές να μας πούν τι προτείνουν. Κύριε Γκυγιόν πρώτα. Σημερίζομαι απόλυτα τη γνώμη του κυρίου Μπουσουτήλ. Μου φαίνεται ότι είναι αδύνατο τέτοιες ώρες να εξετάσουμε ένα θέμα τόσο σημαντικό. Έχουμε ένα σωρό πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Θα έλεγα λοιπόν να αναβάλουμε το θέμα για μια ημερομηνία όπου θα έχουμε περισσότερη ώρα να συζητήσουμε. Η κυρία Βάκστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικός φάκελος αυτός. Και χαίρομαι για την πρόταση που έκανε ο εισηγητής, ο Σάιμον Μπουσάτιλ. Όντω, να αναβάλουμε τη συζήτηση για κάποια άλλη στιγμή, να μπορούν και περισσότεροι συνάδελφοι να είναι παρόντες για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς, η κυρία Κέλλερ. Και εγώ συμφωνώ. Και να είμαστε πιο ρεαλιστικοί όταν φτιάχνουμε ημερήσιες διατάξεις. Νομίζω ότι σήμερα είχαμε βάλει υπερβολικά πολλά θέματα. Είναι προφανές λοιπόν ότι είναι πολύ πιεσμένη η ημερήσια διάταξη. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστούμε. Α, η κυρία Βερζέκη, τώρα το λόγο. Θα σύντομη. Εγώ θα προτιμούσα να είναι ο σκιώδης συγητής της Γκουε που εκφράζεται, αλλά επειδή δεν είναι εδώ, θα πω και εγώ ότι σύμφωνο. Κύριε Μπουσάτελ, εσείς τώρα. Ακούσατε τους σκιώδης εισηγητές και εκπροσώπους της ΛΥΜΠΕ, που είναι πολύ λογικοί και αναγνωρίζουν το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα να συζητήσουμε, τη Frontex. Και γι' αυτό ακριβώς αξίζει περισσότερο χρόνο για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε σήμερα. Μόλις έμαθα ότι η προγραμματισμένη συνάντηση με τους Πολωνούς θα αλλάξει αίθουσα. Συνεπώ, όσοι από εσά θέλουν να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή με την αντιπροσωπεία από την Πολωνική Βουλή, 3Ε2 είναι η αίθουσα όπου έχουμε τη συνάντηση αυτή, η οποία ξεκινάει στις 6.30. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε τον ε, κύριο Μπουσάτιλ τώρα και να φροντίσουμε κάποια άλλη στιγμή να προβλέψουμε την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. γρήγορα βέβαια, στην επόμενη τακτική συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Κύριε Μπουσάτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, από τη μια με απογοητεύει, αλλά από την άλλη μεριά είναι το μόνο λογικό πράγμα να αναβάλουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να επαναλάβω ότι θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι σκιώδες συζητητές να νιώσουν ότι τους δίνουμε αρκετό χρόνο για να μελετήσουν αυτή την υπόθεση. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί τους. Συνεπώς, Πρόεδρε, τώρα ε, προχωράμε, καθυστερούν δηλαδή όλα κατά ένα βήμα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή η προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών όλα τα επόμενα βήματα, όλοι οι επόμενοι σταθμοί στην εξέταση της έκθεσης αυτής θα καθυστερήσουν κατά 15 μέρες. Έτσι δεν είναι. Εγώ θα φροντίσω πάντως την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσω το διάλογο με τους συναδέρφους. Αλλά είναι λογικό και κατά τη γνώμη μου να αναβληθεί το σημείο αυτό. Τέλος, Πρόεδρε. Σας παρακαλώ να φροντίσετε την επόμενη φορά να έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι νομοθετικό ζήτημα, όπως είπα. Άρα έχει μεγάλη σημασία και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να συζητηθεί. Πρόεδρος, βεβαίως κύριε Μπουσούτιλ. Εκτιμάμε όλους ιδιαίτερος την ετοιμότητά σας να αναβάλουμε το ζήτημα αυτό, το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Συμφωνούμε και καλοδεχόμαστε το γεγονός ότι θα συναντηθείτε με τους σκιώδεις εισηγητές την επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη τακτική συνεδρίαση πάντως της ΛΥΜΠΕ θα φροντίσουμε να έχουμε το χρόνο που αξίζει στο θέμα αυτό για να συζητήσουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Και πάλι σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την αναβολή και πάμε στην αίθουσα 3Ε2 για να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους του Πολωνικού Κοινοβουλίου σε μία συνεδρίαση που προβλέπεται για μία ώρα. Σας ευχαριστώ.